Dear colleagues, may you please take seat. Συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε. guest today, but first let's have the agenda adopted. Thank you. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, να εγκρίνουμε πρώτα την ημερήσια διάταξη. Ευχαριστώ. Ανακοινώσει του Πρόεδρου εκτακτή συνεδρίαση την Δευτέρα το βράδυ στο Στρασβούργο. Σχέδιο ημερήσια διάταξη θα το λάβετε σύντομα και θα περιλαμβάνει εξέταση της έκθεση, σχεδίου έκθεσης 2016 καθώς επίσης και συνάντηση με το Ευρωπαϊκό Συμβουλευτικό Όργανο για τα Στατιστικά Στοιχεία. Περνάμε σημείο 3. Καλωσορίζω τον κύριο Μάρκ Κάρνη διοικητή της Τράπεζας Αγγλίας, ε, πρώτο αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Ο κύριος Κάρνη είναι πρώτος αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου από το 2013. Διαδέχτηκε τον Μάρβιν Κίνγκ που είχε την ίδια ιδιότητα ο πρώτος αντιπρόεδρος σύμφωνα με τον κανονισμό που ισχύει πρέπει να παρουσιάσει στο Κοινοβούλιο το πώς σκοπεύει να διεκπαιρεώσει τα καθήκοντά του. Είναι βεβαίως όπως είπαμε διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας, πρέπει όμως να τονίσω ότι σήμερα είναι εδώ πέρα υπό την ιδιότητά του ως πρώτος αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου που εντολή έχει, όπως ξέρετε, την μακροπροληπτική εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ένωσης ε, για να συνεισφέρει στην πρόληψη η μείωση συστημικών κινδύνων ε, στην χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Γι' αυτό σας παρακαλώ να περιοριστούμε σε αυτό το θέμα για το οποίο είναι υπόλογος ο κύριος Κάρνη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βεβαίως ε, το θέμα αυτό από μόνο του είναι και κρίσιμο για την Επιτροπή μας και ευρύτατο οπωσδήποτε. Οπότε οι βουλευτές ε, θα ασχοληθούν με αυτά τα σημαντικά ζητήματα. Λοιπόν, θα ακούσουμε πρώτα την δήλωσή σας και μετά έχουμε πέντε λεπτικές απαντήσεις. Κύριε Διοικητά, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι βουλευτές. Είναι χαρά μου σήμερα το να μπορώ σήμερα να σας μιλήσω ως Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου. Η διατήρηση της ε, χρηματοπιστωτικής σταθερότητας αποτελεί ένα, απαιτεί ένα στεναρό πλαίσιο, ένα, μια αντίληψη του κινδύνου και βεβαίω όπου αυτό είναι αναγκαίο ένα συντονισμό των ε, μακροπροληπτικών πολιτικών. Βεβαίως η ανάγκη του συντονισμού είναι πάρα πολύ σημαντική δεδομένη της μοναδικής φύσης ενιαίας αγοράς και άρα το Συμβούλιο μας προσπαθεί να κάνει την χρηματοπιστωτική πολιτική πιο αποτελεσματική. Τώρα είναι ανοιχτά τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη στηρίζει τον οικονομικό δυναμισμό με το να διευκολύνει το εμπόριο και την εξειδίκευση, το να ενισχύει τον ανταγωνισμό, σημαίνει μεγαλύτερες αγορές, ευρύτερη επιλογή, μεγαλύτερα κίνητρα και οικονομίες κλίμακος. Βεβαίω αυξάνει τον δυναμισμό αλλά αυξάνει και την έκθεση σε σοκ από το εξωτερικό, ειδικά οι χρηματοπιστωτικοί σύνδεσμοι δημιουργούν και νέα ευάλωτα σημεία. Το Συμβουλίο μας λοιπόν μπορεί να βοηθήσει να οικοδομηθεί η απαραίτητη αντοχή έτσι ώστε να ενισχυθούν τα θετικά των ε, ανοιχτών αγορών και να μειωθούν οι κίνδυνοι που αυτό περιέχει. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω τρει σημαντικέ συνεισφορέ που κάναμε όσο εγώ είμαι αντιπρόεδρο. Πρώτα απ' όλα, έχουμε προωθήσει τα στιβαρότερα μακροπροληπτικά πλαίσια. Συγκεκριμένα έχουμε κάνει κάποιες συστάσεις έτσι ώστε οι εθνικοί νομοθέτες να ενισχύσουν αυτό το πλαίσιο στην εθνική νομοθεσία. Έχουμε βγάλει ένα σχετικό εγχειρίδιο το οποίο περιέχει πρακτικές πληροφορίες για το πώς μπορεί να χαραχθεί πολιτική με βάση αυτές τις νέες αρμοδιότητες. Το εγχειρίδιο παρουσιάζει τις βέλτιστες πρακτικές αναμέσω, προτείνει κάποιους δείκτες ε, και καθορίζει και το νομικό πλαίσιο που τα ορίζουν. Επίσης αναφέρει και πιθανές ε, συνέπειες οι οποίες ε, μπορεί να υπάρξουν. Όπου κρίνουμε ότι δεν ακολουθούμε, δεν ακολουθείται η βέλτιστη πρακτική, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το λεγόμενο soft law για να κάνουμε συστάσεις ε, στις οποίες θα πρέπει είτε να συμμορφωθούν είτε να εξηγήσουν τα κράτη-μέλη. Παραδείγματος χάρη, πέρσι, εκτός από κάποιες κατευθυντήριες γραμμές, ακριβώς τις εθνικές μακροπροληπτικές αρχές για να ακολουθήσουν κάποια αντικυκλική πολιτική και το ίδιο θα κάνουμε όσον αφορά και το τρίτο τετράμινο του 2016. Οι τελευταίες μελέτες μας έδειξαν πως ε, υπάρχει ανάγκη να χρησιμοποιηθούν τα περιθώρια που υπάρχουν για να αντιμετωπίστηκε η κύκλικη συμπεριφορά στα παράγωγα και στα αξιόγραφα. Και φέτος βεβαίως ε, σκοπεύσαμε να συμπεριληφθούν ε, τα μακροπροληπτικά περιθώρια στο πλαίσιο ομόχλευσης. Η Τράπεζα της Αγγλίας έχει ακολουθήσει αυτή την προσέγγιση με τρόπο που την καθιστά εύρωστη απέναντι σε κυκλικούς και διαρθρωτικούς κινδύνους. Μια, ένα άλλο ισχυρό σημείο μας είναι η δυνατότητα να συλλέγουμε δεδομένα και να κάνουμε ανάλυση από όλα τα κράτη-μέλη. Όσον αφορά λοιπόν τον λόγο μόχλευσης, συλλέγουμε νέα εμπειρικά δεδομένα που δείχνουν πως η μόχλευση του τραπεζικού τομέα ενίσχυσε τις κυκλικές τάσεις που υπήρχαν σε όλο σχεδόν τα κράτη-μέλη και βλέπουμε πως ο κίνδυνος τίνει να μειώνεται σε επιστοτική επέκταση και να αυξάνεται σε περιόδους ε, ύφεσης. Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή είδαμε πως οι συστημικές τράπεζες ε, στην Ευρώπη έχουν κατά κανόνα πολύ χαμηλό κίνδυνο και ποσοστό μόχλευση σε σχέση με τις άλλες τράπεζες. Ένας άλλος τρόπος με τον οποίο βλέπουμε τις βέλτιστες πρακτικές και επηρεάζουμε το τι γίνεται είναι με το να παίρνουμε μια μακροπροληπτική αντίληψη για το πώς ε, τα στοιχεία του δημοσιονομικού συστήματος μπορούν να επηρεάσουν την μακροχρόνια ευημερία. Παραδείγματο χάρη, εξετάζοντας ε, την οδηγία για την φερικαιότητα 2, βλέπουμε πώς οι μακροπρόθεσμοι επενδυτές όπως τα ασφαλιστικά ταμεία μπορούν να φέρουν μια σταθερότητα στο σύστημα. Κατά την άποψή μας περισσότερα μπορούν να γίνουν στο πλαίσιο της οδηγίας για τη φερεγγιότητα 2 και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συνδημικής Σταθερότητας μπορεί εδώ πέρα να δώσει την σωστή και αντικειμενική προοπτική καθώς το Κοινοβούλιο ετοιμάζεται για μια αναθεώρηση το 2018 και βεβαίω τι αγορές σημαίνει ότι θα πρέπει να αντιλαμβανόμαστε τους ε, κινδύνους. Το Συμβούλιο μας παίζει σημαντικό ρόλο για να αντιληφθούν τα κράτη-μέλη τους ε, νέους κινδύνους. Γνωρίζουμε πως το χρηματοπιστωτικό σύστημα άλλαξε πάρα πολύ από την κρίση σχεδόν όλη η νέα πίστη που δημιουργήθηκε ήταν από τις αγορές ε, ομολόγων και ταυτόχρονα τα στοιχεία ενεργητικού που είναι υποδιαχείριση έχουν αυξηθεί κατά 60% παγκοσμίω και 80% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές οι τάσεις θα συνεχιστούν. Το Συμβούλιο μας λοιπόν συνεισφέρει με δύο τρόπους σε πιο ανθεκτικές ε, κεφαλαιαγορές. αγορέ. Πρώτον, προωθεί μια κοινή αντίληψη των βασικών στοιχείων που ενισχύουν την ρευστότητα και δεύτερον συγκεντρώνει στοιχεία για την φύση και το μέγεθος των κινδύνων που σχετίζονται με το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Ή το Συμβούλιο μας ε, έχει μοναδικές αρμοδιότητες ως προς αυτό και αυτή τη στιγμή ερευνά και τους επέκτες αγοράς και τους διαχειριστές ε, για να δουν το τι θεωρούν ότι μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο στην ε, ρευστότητα της αγοράς. Η έρευνα αυτή θα καταλήξει στο, σε ένα συμπέρασμα για το εάν ε, κάποια ταμεία έχουν επαρκή ρευστότητα για να αντιμετωπίσουν πιθανή ρευστοποίηση στην ε, περίπτωση που η αγορά αντιμετωπίσει κινδύνους. Σε μία ανάλογη έρευνα της ε, Τράπεζας Αγγλίας είδαμε πως υπήρχε σαφώς ένα πρόβλημα όσον αφορά την πιθανή ρευστοποίηση των ε, εταιρικών ομολόγων ε, σε δολάρια. Αναλόγως λοιπόν θα πρέπει να κινηθούμε και όσον αφορά την αντίδρασή μας. Θα γίνουν διάφορα stress test που, τα οποία θα συμπληρώσουν τα υφιστάμενα stress test που υφίστανται οι τράπεζες, οι ασφαλιστικές εταιρείε και τα συνταξιδοτικά ταμεία. Επίσης το Συμβουλίο μας αρχίζει να αξιολογεί τις ε, εκθέσεις που μας δίνουν τα αποθετήρια στα οποία γίνεται το εμπόριο παραγόγων. Με αυτόν τον τρόπο οι αρχές μπορούν καλύτερα να αντιληφθούν το περίπλοκο δίκτυο των συναλλαγών παραγόγων και να δουν πώς μπορεί να ενισχυθεί ή πώς αυξάνεται ο κίνδυνος στο σύστημα. Επίσης μπορούμε να δούμε τι αντίκτυπο θα έχει θα έχουν υποχρεωτικά κεντρικά αποθετήρια. Η τρίτη συνεισφορά που κάνουμε θεωρία του συστήματος είναι να έχουμε κάποιες κοινέ προσεγγίσεις στην ε, διαχείριση του κινδύνου. Σε κάποιες περιπτώσεις οι αρχές δεν αρκεί να καταλαβαίνουν, αλλά θα πρέπει να έχουν και μια κοινή προσέγγιση διαχείρισης ε, του κινδύνου. Το Συμβούλιο μας είναι το μόνο μέρος στο οποίο συγκεντρώνονται όλες οι αρμόδιες αρχές. Οι κεντρικές τράπεζες, οι εποπτικές αρχές, και οι αρχές ε, των χρηματαγορών. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποιες βέλτιστες πρακτικές. Παραδείγματο χάρη όσον αφορά τα ε, ακίνητα και μάλιστα στον τομέα της ε, κατοικίας. Βλέπουμε ακριβώς πώς επηρεάζονται αυτές οι αγορές από τις διαρθρωτικές διαφορές που υπάρχουν, από τους περιορισμούς που υπάρχουν όσον αφορά το ύψος των δανείων σε σχέση με την αξία μέχρι το τι δίνεται ως εγγύηση για να δάνει. τα βασικά μαθήματα που βγαίνουν από την ανάλυση είναι ότι χρειάζεται κάποια ευελιξία όσον αφορά τον σχεδιασμό των μακροπροληπτικών εργαλείων. Δεύτερον, δεν υπάρχει ένα εργαλείο το οποίο θα αντιμετωπίσει όλου του πιθανού κινδύνου. Τρίτον, ότι τα εργαλεία πρέπει βεβαίω να ταιριάζουν με τι συνθήκε τη κάθε χώρα. Και τρίτον, πω οι εγχώριε πολιτικέ είναι πιο αποτελεσματικέ και για την εγχώρια και για την ευρωπαϊκή σταθερότητα. Το Συμβούλιο μας λοιπόν έχει οικοδομήσει ένα πλαίσιο για την διαχείριση της διάχυσης αυτού του κινδύνου, το οποίο νομίζω θα συμφωνήσουμε αρχές του επομένου έτους. Το βασικό του στοιχείο είναι η αμοιβαιότητα, να μην υπάρχει δηλαδή το ρυθμιστικό αρπιτράζ, έτσι ώστε να έχει μεγαλύτερη ισχύ η εγχώρια νομοθεσία. Θα βασιστούμε λοιπόν κυρίω στι συστάσει του Συμβουλίου μα και θα πρέπει τα κάτι μέλη να συμμορφωθούν και να εξηγήσουν γιατί δεν συμμορφώνονται. Και βεβαίω ε, ενημερωθήκαμε για μακροπροληπτικές ε, δράσει, 69 φορέ ε, πέρσι και 173 φορέ από όταν υιοθετήθηκε η οδηγία για την κεφαλαιακή επάρκεια το 2014. Παρά το ότι πολλά από αυτά είναι τελείω διαδικαστικά, δείχνουν τι γενικότερε κατευθύνσει. Πάρα πολλέ χώρε χρησιμοποιούν μακροπροληπτικά εργαλεία. Επίση, το Συμβούλιο μας ε, θα αξιολογήσει το πώς οι εθνικές μακροπροληπτικές αρχές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα αποθέματα κεφαλαίων για να κάνουν αντικυκλική πολιτική από χώρε και εκτός της ε, ΕΟΧ. Κάτι το οποίο μας δίνεται από το δίκαιο το οποίο μας διέπει. Και ενώ βεβαίω οι κίνδυνοι στον τομέα των ακινήτων απορρέουν από εθνικές διαφορές, κάποιοι άλλοι κίνδυνοι απορρέουν από λανθασμένη συμπεριφορά. Τα τελευταία χρόνια τα πρόστιμα που επιβάλαμε είναι πάνω από 50 δισεκατομμύρια ευρώ, κάτι το οποίο έχει άμεσες επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία. Με ένα ποσοστό του 5% το κεφάλαιο αυτό θα μπορούσε να είχε υποστηρίξει 1 τρισεκατομμύριο ευρώ σε δάνεια. Επιπλέον, όταν έχουμε επανειλημμένα επεισόδια, υπονομεύεται η πίστη του κοινού στο σύστημα. Οπότε, σκοπεύουμε να ανοικοδομήσουμε αυτή την εμπιστοσύνη. Πρώτα απ' όλα, σκοπεύουμε να συμπεριλάβουμε το κόστος των προστήμων στα stress test. Και η Τράπεζα της Αγγλίας ε, έχει ακολουθήσει αυτή την συμβουλή και έχουμε συμπεριλάβει άλλα 40 δισεκατομμύρια λίρες ε, όσον αφορά το κόστος μη συμμόρφωσης επιπλέον προτείναμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα στην πηγή του με το να αυξήσουμε την λογοδοσία. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω της ε, μεταρρύθμισης ε, των αμοιβών, οι οποίες θα πρέπει να είναι κειμενόμενες και θα συνδυάζονται με ένα σύστημα μάλους, ε, καθώς και ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων. κάτι για το οποίο έχει δεσμευτεί το Ηνωμένο Βασίλειο. Όμως η αποτελεσματικότητα αυτών των μέτρων βεβαίως περιορίζεται και από το πλαφόν που υπάρχει στα μπόνους. Παραδείγματος χάρη, το 2013 στις μεγάλες τράπεζες του Ηνωμένου Βασιλείου ο λόγος μεταξύ σταθερής ε, και μη αμοιβή ήταν γύρω στο 1 προς 3. Δηλαδή τα 3 τέταρτα των αμοιβών κινδύνευαν εάν υπήρχε κάποια λανθασμένη συμπεριφορά. Να με συγχωρείτε, μιλούσα λίγο γρήγορα για να προλάβω το χρόνο. Και βεβαίω ε, το 2014 όταν έπρεπε να εφαρμοστεί το πλαφόν στα μπόνους, ο λόγος αυτός μειώθηκε στο 1 προς 1. Ενώ το συνολικό επίπεδο αμοιβών έμεινε ανεπηρέαστο. Με την παρακίνηση του Συμβουλίου μας, το Συμβούλιο Δημοσιονομικής Σταθερότητας τώρα εξετάζει το πώς επηρεάζουν τα διάφορα μοντέλα αμοιβών την ε, λανθασμένη συμπεριφορά και θα κάνει συστάσεις ε, στην επόμενη σύνοδο των ε, G20. Βεβαίω οι συστάσεις είναι αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη. Θα πρέπει να γίνουν περισσότερα για να λογοδοτούν τα άτομα. Εν μέρη λοιπόν, χάρη στην παρακίνηση του Συμβουλίου μας, το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα μοιραστεί τις εμπειρίες του για τον ρόλο των ρυθμιστικών ε, αρμοδιοτήτων των ε, τραπεζών για να αντιμετωπίσουν ακριβώς τέτοιες ε, συμπεριφορές. Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε ένα νέο καθεστώς έτσι ώστε η διοίκηση σε διάφορους οργανισμούς να είναι απευθείας και ατομικά υπεύθυνη για τους τομείς αρμοδιότητάς τους, κάτι το οποίο βεβαίως θα συνοδευτεί και από έναν κώδικα συμπεριφοράς έτσι ώστε να γίνουν αυτά αντιληπτά από όλους. Συμπερασματικά λοιπόν, όλα τα κράτη-μέλη και βεβαίως όπως ξέρετε οι πολίτες της Ένωσης ε, έχουν ένα συμφέρον προς την, ε, με την δημοσιονομική σταθερότητα. Και βεβαίως η κρίση κατέδειξε πόσο γρήγορα μπορεί να διασχίσει τα σύνορα ο κίνδυνος και άρα θα πρέπει να υπάρξουν ε, μεταρρυθμίσεις και μια νέα προσέγγιση με την ηγεσία που επιδεικνύει η Επιτροπή σας το πρόγραμμα αυτό των μεταρρυθμίσεων ουσιαστικά έχει ολοκληρωθεί και οι αρχές πλέον τώρα εστιάζουν στο να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά του. Αλλά η σταθερότητα απαιτεί κάτι περισσότερο από μακροπροληπτικά μέτρα για να αντέξουν μεμονωμένες εταιρείες. Απαιτεί μια μακροπροληπτική λογική με την ευελιξία για να μπορούμε να αντιδρούμε σε σοκ όπου και αυτά εμφανιστούν με υψηλότερες και αυστηρότερες προταγραφές για τις συστημικά σημαντικές εταιρείες. Το Συμβουλίο μας βοηθά τα κρατημέλη να εκπληρώσουν αυτούς τους ρόλους και βεβαίως παρακολουθεί και τις νέες αδυναμίες όπως περιέγραψε πρόσφατα και ο πρόεδρος Ντράγκη τα επόμενα έτη το Συμβούλιο μας θα αξιολογήσει την μακροπροληπτική στάση των κρατών μελών για να συμπληρώσει την παρακολούθηση του κινδύνου και θα δει τους κινδύνους των χαμηλών επιτεκείων στην ε, χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την απότομη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλή άνθρωπη. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Ευχαριστούμε κύριε Κάρνη ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η παρέμβασή σας και καλύψατε ένα ευρύ φάσμα σημαντικών ε, για μας ζητημάτων για τα επενδυτικά ταμεία, για την, ε, το υποχρεωτικό clearing, ε, για το ανώτατο όριο των πόνους, για την αποτίμηση της μακροληπτικής ε, θέσης που υιοθετούν τα κράτη-μέλη. Σίγουρα θα είναι συνταρακτική η συζήτηση που θα κάνουμε. Ε, ας ακούσουμε τους προσώπους πολιτικών ομάδων, κύριος Κύριε Διοικητά, θα μιλήσω γερμανικά. Πρώτα απ' όλα, σας ευχαριστώ που ήρθατε στην Επιτροπή μας. Το εκτιμούμε και σας γνωρίζουμε βεβαίως από την μεταβατική φάση προεδρία σας. Αλλά βεβαίως αυτό πέρασε και ορίστηκε ξανά ο Μάριο Ντραγκή. Λοιπόν, έχω δύο ερωτήσεις ε, κύριε Διοικητά. Πρώτα απ' όλα γνωρίζετε τις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις ε, στον τομέα της νομοθεσίας ε, μόλις μας το είπατε και πριν από λίγες εβδομάδες ε, στην Ατάλια στην Τουρκία είχαμε την σύνοδο των G20 και εκεί πέρα αναφέρθηκε και αποφασίστηκε μία νέα προδιαγραφή τη λέξη για τις συστημικά σημαντικές τράπεζες και Έχουμε επίσης ε, και από το δικό σας σύστημα νομικά δεσμευτικά αποθέματα απολειών με το λεγόμενο υπορδιαγραφή Embrae. Θα ήθελα λοιπόν ε, να μου πείτε αν θα πρέπει να υπάρχει σύντομα ένα ποσοτικό τέτοιο υποχρεωτικό προδιαγραφής ε, γύρω στο 8% του ισολογισμού και πώς ε, οι δύο πρωτεγραφές Έμπρεϊ και Τίλαγκ θα μπορούν να λειτουργήσουν από κοινού. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε παράταση του προγράμματος αγοράς αξιογράφων. Η ρευστότητα στον τραπεζικό τομέα είναι πάρα πολύ υψηλή εδώ και καιρό, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει οδηγήσει σε βελτίωση των ε, επενδύσεων ανταυτού. Οι τράπεζες και ασφαλιστικές ε, εταιρείε ε, προτιμούν πιο επικερδείς επενδύσεις. Ε, θα ήθελα λοιπόν να μάθω πώς αξιολογείτε εσείς πέρα από αυτά τα οποία μας είπατε τον ε, συστημικό κίνδυνο στο χρηματοπιστωτικό τομέα, ειδικά όσον αφορά τον κλάδο των ασφαλιών. Ευχαριστώ. Um, Ευχαριστώ. Πολύ σημαντικές και οι δύο ερωτήσεις. Το ξέρω ότι το ξέρετε, αλλά θα ήθελα να διευκρινίσω για το TILAC, που ενέκριναν, το πρότυπο που ενέκρινε ε, η G20 είναι το πρότυπο που ισχύει για τις 20 μεγαλύτερες συστημικά σημαντικές τράπεζες και έπρεπε να συμφωνηθεί ανά τον κόσμο από τη ΣΥΠΑ μέχρι την Κίνα από όλες τις συναρμόδιες αρχές και ο στόχος ήταν να παράσχει αυξημένη εμπιστοσύνη για εξαιρετικά ε, περίπλοκες διασυνοριακές οντότητες και γι' αυτό το τίλαξε είναι πιο πρόσφορο σε σχέση με το Emerald ε, είναι ε, μια ευρύτερη αν θέλετε δομή και για να γίνει πιο αυτό, αυτό που λέω θα σας εξηγήσω ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε συστημικά σημαντικές ε, τράπεζες και εσείς το ίδιο στη χώρα σας. Το T-Lag θα το εφαρμόσουμε μέσω του Emerald και Το έγγραφό μας για την εφαρμογή του θα δημοσιοποιηθεί στις αρχές του Ιανουαρίου και θα δώσει περισσότερες λεπτομέρειες και φυσικά όπως καταλαβαίνετε θα καλύψουμε ένα ευρύτερο φάσμα ε, θεσμών ε, οντοτήτων ε, ανάλογα με, το, με τη συστημική του σημασία. Το βασικό στοιχείο που θα ήθελα να τονίσω για να περάσω ταχύτερα και στη δεύτερη ερώτησή σας, διότι δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Δεν μιλάμε μόνο για την μειωμένη ικανότητα απορρόφησης που θα δημιουργηθεί μέσα του Emerald ή του τιλεκ αλλά η γνώση του ότι υπάγονται σε κανόνες αυτά τα όργανα και άρα υπάρχει μεγαλύτερη ρύθμιση, μεγαλύτερη πειθαρχία, δηλαδή Κανονικά θα έπρεπε αυτοί που έχουν το κεφάλαιο να ε, υπάγονται σε αυτή την πειθαρχία, όμως δεν συνέβη αυτό και γι' αυτό έχουμε αυτή την πυραμίδα, αν θέλετε, πειθαρχία μέσω των κανόνων. Και τώρα, ε, ε, για την νομισματική πολιτική, αυτή τη στιγμή είμαι σε, σε εφεδρεία αν θέλετε δεν ασχολούμαι αλλά παρόλα αυτά θα σας έλεγα ότι σε συνεργασία με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ασχολούμαστε με την σύνθεση του χαρτοφυλακίου, δηλαδή για, θέλουμε να περάσουν οι επενδυτές σε νέες μορφές επενδύσεων όπως τα ομόλογα της Ιταλικής κυβέρνησης. Τους πιέζουμε σε αυξημένο κίνδυνο, σε αλλοδαπά δηλαδή στοιχεία ενεργητικού και γι' αυτό περνάμε και από τις ισοτιμίες, από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Σας ευχαριστούμε η Ελίζα Φερέιρα. Θα τα πω στα αγγλικά. για να διευκολύνω την επικοινωνία. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Θα ήθελα να επανέλθω στις αρχές του ESRB. Ε, εξ αρχής δεσμεύτηκε το Κοινοβούλιο και ε, με διορθώσει και ο συνάδελφος διότι ήταν εισηγητής μαζί με τη Σίλβια Γκουλάρ για αυτό το θέμα. Εξ αρχής προσπαθούσαμε να έχουμε μια σφαιρική εικόνα και να μην ασχολούμαστε με τις μεμονωμένες λεπτομέρειες, τόσο ώστε να πραγματευόμαστε πραγματικά το συστημικό κίνδυνο στην Ευρώπη. Αναρωτιέμαι, σε σχέση ε, με αυτό το τελευταίο κομμάτι της ε, παρέμβασή σας για την ε, μακροληπτική εποπτεία. Πώς θα λειτουργήσει αυτό στην Ευρώπη κατά τη γνώμη σας, ε, διότι έχουμε την ποσοτική χαλάρωση ε, και πώς θα συνδυαστεί με την μακροληπτική εποπτεία στο βαθμό που δεν ανταποκρίνεται στην ποσοτική χαλάρωση η πραγματική οικονομία και επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικό, έχετε την εμπειρία από το Ηνωμένο Βασίλειο, από τη ΣΥΠΑ, από τον Καναδά, τι λείπει, ποιο συστατικό λείπει από το ευρωπαϊκό μίξ για να λειτουργήσει αυτή η προσπάθεια Δεύτερον, ε, αυτή τη στιγμή ασχολούμαστε ναι, με, με την ε, Κεφαλαϊκή Ένωση, αλλά ακόμη και χωρίς νέα νομοθεσία δεν λειτουργεί, δεν η Τραπεζική Ένωση, διότι λείπουν σκέλη. Το δεύτερο, το τρίτο, ε, σκέλος δεν λειτουργούν, λείπουν στοιχεία και είναι πολύ περίεργο να περάσουμε σε ένα νέο εγχείρημα πρωτού ολοκληρώσουμε το προηγούμενο. Και τρίτον, το ο ευρωπαϊκός ε, συστημικός κίνδυνος ε, ή ας το πω αλλιώς ε, θα συμμετάσχει ή όχι το Ηνωμένο Βασίλειο. Ζητώ συγγνώμη σας θέτω αυτό το ερώτημα, αλλά είναι αναπόφευκτο. Ήρθατε εδώ και πρέπει να το θέσω ανοιχτά αυτό το ερώτημα. Και φυσικά θα απαντήσετε στο μέτρο που επιθυμείτε, αλλά είναι θέμα Ε, υπάρχει ε, συστημικός κίνδυνος ή συστημική ευκαιρία για το ε, κοινό νόμισμα. Απάντηση. Εξαιρετικές ερωτήσεις. Θα αρχίσω με την πρώτη. Το περιβάλλον κινδύνου. Δεν είναι μοναδικό χαρακτηριστικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε όλες τις προηγμένες σας πω έτσι όπου υπάρχουν υπάρχουν ε, διαφορετικές ε, πορείες ε, ναι μεν για την νομισματική πολιτική όμως βασιζόμαστε μετά την κρίση στην δυνατότητα δανειοληψίας και Συνδυάζοντας αυτό με τις δημογραφικές εξελίξεις, ε, τις κεφαλογικές απαιτήσεις και τη δανειοληπτική ε, και δανειοδοτική ικανότητα, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες να έχουμε χαμηλότερες ε, πιθανότητες να το πετύχουμε σε σχέση με το παρελθόν και εξάλλου αυτό εξαρτάται και από την τιμολόγηση των στοιχείων του ενεργητικού. Υφίσταται κίνδυνος και φυσικά ελοχεύει πάντοτε αυτός ο κίνδυνος σε κομμάτια πραγματικών οικονομιών να δημιουργηθεί αυτός ο κίνδυνος και γι' αυτό χρειαζόμαστε την στρατηγική μακροληπτικής εποπτείας. Έχουμε διαφορετικές δομές μέσα σε κάθε οικονομία και άρα ε, στα, στο τομέα των ακινήτων μπορεί να εμφανιστεί η κρίση σε εμπορικό επίπεδο ή επίπεδο ιδιωτών και γι' αυτό περνάω στο δεύτερο, στη δεύτερη δέσμη ερωτημάτων, που σχετίζονται με τα οικονομικά, που σχετίζονται με την αγορά. Δηλαδή πώς μπορείτε να επιτύχετε Είχετε τη διαφοροποίηση, την ποικιλομορφία και άρα και την αθεκνικότητα μέσα σε μια αγορά, μέσα από την τιτλοποίηση. Όπως σας είπα και στις αρχικές παρατηρήσεις, η συμμετοχή πιο μακροπρόθεσμων επενδυτών όπως ε, οι ασφαλιστικές εταιρείες ε, προϋποθέτει ότι ε, θα έχουμε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων στις κεφαλαίες αγορές. Αυτό είναι καθοριστική σημασία όχι μόνο για να αυξήσουμε, να είναι πιο εύρωστη η οικονομία αλλά και πιο ανθεκτική. Για τις ερωτήσεις για την Τραπεζική Ένωση μπορώ ακροφυγούς μόνο να αναφερθώ στο ζήτημα αυτό, υποθέτω πως ε, από τη δική μου τη σκοπιά θεωρώ ότι χρειαζόμαστε και τα δύο, και την κεφαλαιοκή και την τραπεζική ένωση. Χρειαζόμαστε και τα, τις δύο αυτές διαστάσεις, ούτως ώστε να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε την θεσμική δομή Τη ε, οικονομία και να προωθήσουμε την Τραπεζική Ένωση φυσικά με τον πλέον ε, ε πρόσφορο τρόπο, αλλά ε, καθοριστική σημασία είναι να συνεχίσουμε τι προσπάθειες. Αυτή τη στιγμή η Τραπεζική Ένωση είναι, αν θέλετε, ένα σταθμό στο ταξίδι που κάνουμε και η συνέπεια είναι ότι θα υπάρξουν κίνδυνοι στο βαθμό που ενδεχομένως μπορούν να ανακύψουν εξωγενή σοκ για τις οικονομίες. Τώρα, αυτό που με ρωτήσατε για το Ηνωμένο Βασίλειο και τη σχέση του με το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν ε, συμμετέχω καθόλου στις ε, συζητήσεις ε, Brexit. Το... Ο στόχος είναι να παίρνουμε το σύστημα της Ευρωπαϊκή όπω είναι και να συνεργαζόμαστε μαζί του. Κάποιοι θέλουν να το κάνουν πιο αποτελεσματικό. Συνεχίζουμε να μαθαίνουμε και να αναπτύσσουμε τις γνώσει και ικανότητέ μα που έχουμε για την μακροληπτική εποπτεία. Στο θέσω έτσι. Καταπληκτική η απάντηση για το ζήτημα. Ευχαριστούμε. Ε, Ευχαριστώ. Εγώ έχω μια ερώτηση που επικαλύπτει δύο συστήματα νομοθεσίας που προσπαθεί να τοποθετήσει τα προϊόντα στην αγορά των παραγωγών αλλά και στην τραπεζαγορά. Έχουμε μια οδηγία σύμφωνα με την οποία είναι εφικτή η σύγκληση μεταξύ των διαφόρων προϊόντων και έχουμε και τη CRD 4. Ωστόσο, ο υπολογισμό τη Βασιλεία 3 και το πώ αυτό το ερμηνεύουμε μέσα στο πλαίσιο του CRD4, απαιτούμε ε, να υπάρχουν περιθώρια αρχικά υποχρεωτικά όσον αφορά τι καταθέσει. Αυτά τα περιθώρια δεν είναι ε, άμεσα ευθύνη των πελατών, είναι ε, αντίστοιχα με το CCP4. Ήδη ορισμένα μέλη καθαρίσεων έχουν σταματήσει να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε κάποιους πελάτες και κάποιοι άλλοι περιορίζουν την έκθεσή τους. Φαίνεται ότι υπάρχει μια αυτόματη προσαρμογή. Όσοι συμφωνείτε πως αυτά τα πράγματα αλλάζουν και αν ναι, εάν η Επιτροπή της Βασιλείας δεν μπορέσει να συμφωνήσει, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δράσει μονομερός. Σας ευχαριστώ πολύ. Να σας πω εξ Εμείς ε, επικροτούμε την προσέγγιση της κεντρικής εκαθάρισης. Αυτό σίγουρα αποτελεί ενίσχυση της κεντρικής αντοχής του συστήματος διότι οι σχέσεις των παραγωγών δεν μπορούσαν να ρυθμιστούν σε κανονικές συνθήκες, πόσο μάλλον σε συνθήκες ε, σοκ. Ε, οι κεντρικοί εκαθαριστές ήδη είναι ολοένα ε, και περισσότερο συστημικοί λόγω του, της κεντρικής φύσης του συστήματος και μπορούμε εκεί να λύσουμε τα προβλήματα πιο εύκολα. Εμείς έχουμε περάσει πολύ χρόνο στον σχεδιασμό σε διεθνέ επίπεδο, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν τα κατάλληλα κίνητρα για τους ε, θεσμούς να εκαθαρίζουν κεντρικά και να μην έχουν διμερές εμπόριο. Ε, ούτε διμερείς απαιτήσει ε, αποθεμάτων ή περιθωρίων. Αυτό μπορεί να τυποποιηθεί έτσι ώστε η κεντρική καθάριση να αποφέρει οικονομίες κλίμακας περιλαμβανομένες και της ανθεκτικότητας αλλά και να αποφεύγονται και οι διμερείς επαφές και εμπόρειες. Σε αυτή τη διαδικασία ωστόσο θα πρέπει να αναγνωρίσουμε και εδώ κινούμε προς την απάντηση της ερώτησής ότι υπάρχουν οικονομίες κλίμακας όχι μόνο για το κεντρικό καθαριστή αλλά και για την τράπεζα αν θέλετε ή το οργανισμό που προβαίνει στην εκαθάριση των παραγόγων. Είναι καλύτερο από το να έχει ένα ευρύτερο χαρτοφυλάκιο παραγόγων ή αξιογράφων. Αυτό σημαίνει ότι άλλοι θεσμοί εξαρτώνται από το ίδιο καθαριστικό σύστημα και αυτό ακριβώς απαντά στη δική σας ερώτηση. Δηλαδή, αν το μοχλευμένο, μοχλευμένη αναλογία περιορίζει την παροχή ε, υπηρεσίας προς τον έμεσο εκαθαριστή, του δεν έχουμε τα πλήρη ωφέλη του συστήματος. Δίνουμε περισσότερα κίνητρα για μεγαλύτερη συγκέντρωση της, ε, σε των συναλλαγών άμεσα μέσω αυτών των μεγάλων εκαθαριστικών κέντρων, έτσι ώστε να περιορίζει το χρόνο, η διαφοροποίηση και η χρηματοπιστωτική σταθερότητα για το σύστημα. Ενώ αν κάνουμε ένα βήμα πίσω, δεν είναι πολύ ε- έξυπνο αυτό για τη διαχείριση του συστήματος. Δεν είναι ο καλύτερος τρόπος διαχείρισης του. Και όταν αρχικά σχεδιάσαμε αυτό το σύστημα στην Ευρώπη, ακολουθήσαμε μια όσο γίνεται πιο ολιστική άποψη του συστήματος ώστε να δώσουμε περισσότερα κίνητρα. Το θέμα είναι κατά πόσο χρειάζεται να προσαρμοστεί η αναλογία μόχλευσης. Δυστυχώς όπως γνωρίζετε είναι μια απέτηση ε, αποκάλυψης και όχι δεσμευτική, ε, δεσμευτική ρυθμιστική απέτηση. Θα πρέπει να υπάρξει ευρωπαϊκή διαδικασία ώστε να ληφθεί απόφαση για αυτό το θέμα. Νομίζω πως αυτό θα πρέπει να είναι πρώτης προτεραιότητας θέμα που θα πρέπει να εξεταστεί όταν θα αποφασίσει η Ευρώπη για εφαρμογή της αναλογίας μόχλευσης. Όμως θα πρέπει να εξασφαλίσουμε πως αυτό δεν θα οδηγήσει σε περίτη αύξηση της αναλογίας μόχλευσης. Υπάρχουν ε, ορισμένες ε, συνέπειες της νομοθεσίας αυτής, ε, οι οποίες δεν ήταν επιθυμητές εξ αρχής σε διεθνές επίπεδο και αυτό θα πρέπει να τη λάβουμε υπόψη μέσω της κατάλληλης διαδικασίας της Βασιλείας, αλλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, άσχετα από αυτό, θα πρέπει να το λάβουμε και εκεί υπόψη. Τέλος, το θέμα αυτό φαίνεται να είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη ΣΥΠΑ λόγω του συμπληρωματικού, συμπληρωματικής αναλογίας μόχλευσης που εφαρμόζεται για τους μεγαλύτερους εμπόρους παραγόγων, τον ΙΠΑ. Ευχαριστώ, η Σιλβί Γκουλάρ. Σας ευχαριστώ, κύριε Δικητά. Είμαι ευτυχή που είστε εδώ γιατί είναι καταρχήν σημαντικό να γίνεται τέτοιο είδου διάλογο και έπειτα γιατί δυστυχώ για εσά ήμουν και ο, η συγγήτρια για το νομοσχέδιο τη ΕΖΑ. Έχω δύο ερωτήσει, ε, λοιπόν. Ε, ε, θεωρείτε πω αυτό ο οργανισμό είναι αρκετά καλά εξοπλισμένο, ώστε να ενισχύσει την ευρωπαϊκή φωνή στις διεθνείς διαπραγματεύσεις γιατί το πρόβλημα που είχαμε ήταν να επιτρέψουμε στην Ευρώπη να κρατήσει τη σειρά και να μπορεί να εκφραστεί σε παγκόσμια επίπεδο. Και το ο κύριος Μπάλτς το ανέφερε και το τίλακ για τις ασφαλίσεις. Υπάρχουν διάφορα που γίνονται και τα οποία επηρεάζονται και από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και μπορεί να είναι πολύ σημαντικά. Και δεύτερον, μήπως είστε εξαιρετικά πολύ στο Συμβούλιο αυτό, σε αυτή την Επιτροπή μάλλον Συστημικού Κινδύνου. Γιατί όταν δημιουργήθηκε αυτό είχαμε κάποιες αμφιβολίες, αλλά δεν ήταν δυνατόν να αλλάξουμε όλες τις διατάξεις, αλλά από την πράξη ρεαλιστικά. Πιστεύετε πως θα έπρεπε κάπως να μειωθεί ο αριθμός των συμμετεχόντων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Εγώ θα σας απαντήσω στα αγγλικά, αν δεν σας πειράζει. Νομίζω πως το θέμα της μεγιστοποίησης του αντικτύπου του Συμβουλίου ε, σε διεθνές επίπεδο θα σας απαντήσω ότι υπάρχουν δύο τρόποι για να το κάνουμε αυτό. Να πάρουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα σε ένα από τα οποία αναφέρθηκα στις αρχικές μου παρατηρήσεις, δηλαδή μοναδική του δυνατότητα να συλλέγει στοιχεία από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τη μεγαλύτερη δηλαδή οικονομία του κόσμου και το μεγαλύτερο οικονομικό σύστημα του κόσμου. Αλλά για να μπορεί να το κάνει αυτό, θα πρέπει να δούμε ότι θα πρέπει να γίνεται το ίδιο και στις υπόλοιπες μεγάλες οικονομίες, όπως τις είπα, όπου ορισμένες φορές ε, δεν μιλούν όλοι μεταξύ τους στον ίδιο βαθμό, ούτε μοιράζονται τα στοιχεία μεταξύ τους τόσο γρήγορα και τόσο αποτελεσματικά. Και στον Καναδά, στη χώρα μου, παλεύουμε με αυτό το θέμα λόγω ακριβώς των διαφορετικών επιπέδων ευθύνης. Αυτές οι αρμοδιότητες μπορούν να χρησιμοποιηθούν λοιπόν και να γίνει ανάλυση με βάση τα στοιχεία και αυτό είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό. Και εμείς ως μέλη του SRB πρέπει αυτό να το χρησιμοποιήσουμε όσο γίνεται περισσότερο. Φυσικά επίσης πρέπει να εστιάσουμε, να εστιάσουμε στα πιο σημαντικά θέματα για την Ευρώπη και κατ' επέκταση και διεθνώς. με βάση μια ανάλυση κινδύνου η οποία να είναι άμεση αλλά να ε, βασίζεται και στο μέσο πρόθεσμο πεδίο και που θα συγκεντρώνει τις διάφορες ε, ε, μεταρρυθμιστικές αλλαγές, θα συνδυάζει τις αλλαγές, θα βρίσκει τους τομείς που ίσως έχουν ξεφύγει και θα μπορεί να τα συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία. Τώρα όσον αφορά τη μεγιστοποίηση του αντικτύπου είναι αρκετά χρήσιμες οι εκθέσεις ε, της ESRB τις οποίες ε, χρησιμοποιούμε και εμείς ε, τις εκθέσεις δηλαδή του Ντράγκη που χρησιμεύουν για να προχωρήσει η συζήτηση κάθε φορά. Είμαστε πάρα πολλοί. Είμαστε υπερβολικά πολλοί. Είμαστε πολλοί και στην ε, FSP. Έχουμε περιφερειακές ομάδες και μέσω των περιφερειακών ομάδων φτάνουμε τους 150 περίπου. Δεν είναι επίσημα πλήρη μέλη, αλλά μέσω αυτών των ομάδων ε, γίνεται η συνεννόηση. Έχουμε τη Διοικητική Επιτροπή. όπου συνεδριάζουμε τακτικά, κάνουμε και τηλεδιασκέψεις και αυτός είναι ένας μηχανισμός ώστε να γίνεται βαθύτερα ο διάλογος για αυτά τα τόσο περίπλοκα ζητήματα. Και μετά υπάρχουν και συγκεκριμένα οδοί εργασίας όπου εργάζονται ανώτατοι υπάλληλοι και νομίζω πως αυτή είναι μια κατεύθυνση την οποία θα πρέπει να ακολουθήσουμε ώστε να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε όσο γίνεται περισσότερο την μεγάλη εμπειρία που έχουν όλοι αυτοί οι συνάδελφοι στην Φραγκφούρτη. Ευχαριστώ ο Φίλιπ Λάμπερτς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε κύριε Δικητά. Τώρα είμαστε στο ίμιση της COP21 και δεν θα σας ε, ε, εκπλήξει ότι θέλω να σας ρωτήσω ε, τη γνώμη σας στη συνέχεια των παρατηρήσεών σας του Σεπτεμβρίου όσον αφορά την χρήση διαφόρων ε, αξιών που έχουμε. Το θέμα είναι για εμάς τι πρέπει να κάνουμε. Εμείς μπορούμε να βλέπουμε τον κίνδυνο, μπορούμε και να τον μετράμε, αλλά κάτι πρέπει να κάνουμε. Και εδώ ακριβώς είδα ότι οι παρατηρήσεις σας ήταν λίγο ελλειπείς, με την έννοια ότι εσείς υποστηρίζετε την ε, εθελούσια, έναν μηχανισμό εθελούσιας αποκάλυψης, αλλά πιστεύετε πως αυτό αρκεί ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτόν τον κίνδυνο, γιατί φαντάζομαι πως ίσως να, να χρειαστούν και πιο δυνατά μέσα, αλλά από ό,τι κατάλαβα εσείς δεν πιστεύετε ότι θα πρέπει η νομοθεσία να αντιμετωπίσει αυτό το κίνδυνο. Πώς μπορούμε λοιπόν να ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο ε, χρηματοπιστωτικής αστάθειας που συνδέεται με τις κλιματικές αλλαγές. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Όπως ξέρετε, στην ομιλία μου εκείνη είχα φέρει το επιχείρημα ότι με την εξαίρεση του κλάδου των ασφαλιών, των αντασφαλιών, οι βασικοί κίνδυνοι της κλιματικής αλλαγής δεν ε, επηρεάζουν τον πυρήνα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Δηλαδή δεν εννοείται και ότι πρέπει να δούμε παραδείγματος χάρη την προληπτική νομοθεσία για να αλλάξει το πώς ε, αξιολογούνται τα δάνεια σε κάποιες επιχειρήσεις ε, λόγω κλιματικού κινδύνου. Γιατί οι κίνδυνοι αυτοί θα εκδηλωθούν όπως λέμε εμείς πέρα από τον ορίζοντα, σε βάθος χρόνου. Οπότε λογικό τρόπο αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων είναι κάποιε υποχρεώσει ε, δημοσιότητα. δεδομένου του ότι όπω είπατε μεγάλο κίνδυνος είναι η μετάβαση προ μια οικονομία χαμηλού άνθρακα. Μια μετάβαση η οποία θα επηρεαστεί από κοινοβούλια, αυτό εδώ το κοινοβούλιο, από κοινοβούλια σε όλο τον κόσμο που θα λάβουν αποφάσεις για την πορεία αυτή μέσω διαφόρων κανονισμών, μηχανισμών για να διαχειριστούν ακριβώς αυτή τη μετάβαση και βεβαίω θα επηρεαστεί και θα καθοριστεί τελικά από την ιδιωτική πρωτοβουλία όσον αφορά την τεχνολογία, την καινοτομία κτλ. Η αξία της ε, δημοσιότητας ε, είναι δυτή. Και οπωσδήποτε η ομάδα εργασίας που έχει συστήσει τώρα το Συμβούλιο Συνδικής Σταθερότητας υπό την Προεδρία του Μάικλ Bloomberg θα είναι λοιπόν του ιδιωτικού τομέα. Θα έχει αυτούς που εκδίδουν ε, αξιόγραφα, αυτούς που παρέχουν κεφάλαια κτλ. για να έχουμε κάποια πράγματα τα οποία θα είναι ξεκάθαρα συγκρίσιμα και αποτελεσματικά. Και θα σέβονται οπωσδήποτε την αρχή της αναλογικότητας και της σημαντικότητας. Η αξία λοιπόν είναι δυτή. Το ένα είναι ότι μας δίνει την απάντηση σήμερα όσον αφορά το αποτύπωμα αερίων θερμοκηπίου των εταιριών, κάτι το οποίο μπορεί να είναι προφανές στις εξορρυκτικές εταιρείε, αλλά δεν είναι τόσο προφανές ε, για ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή για μια εταιρεία πληροφορικής. Τα ξέρετε αυτά φαντάζομαι. Υπάρχουν διάφορες μελέτες ότι, που δείχνουν ότι δεν είναι συγκρίσιμα αυτά τα πράγματα, οπότε για να υπάρχει μια συνέπεια και μια συγκρισιμότητα, ε, ήδη αυτό έχει μια αξία, αλλά και αυτό το οποίο μπορούμε επίσης να ρωτήσουμε είναι ποια είναι η στρατηγική της καφετερίας για να μειωθεί αυτό το αποτύπωμα και σε πιο βάθος χρόνου. Και αυτό μπορεί να γίνει με διάφορους ε, τρόπους. Αυτό θα το κρίνει βεβαίως αυτή η task force, αλλά τώρα το εάν αυτό βασίζεται σε εθνική συνεισφορά της κάθε χώρας. Ναι, ναι, σας ευχαριστώ. Τη συνεισφορά, όπως είπατε για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι γύρω στο 1,5% της 100 ε, μείωση κάθε χρόνο. Το αν μια εταιρεία κινείται προς αυτή την τάξη μεγέθους ή αν δεν κινείται γιατί όχι, είναι ένας μηχανισμός εφαρμογής. Και εάν στο COP21 έχουμε μια επιτυχία, βλέπουμε πως υπάρχει και προοπτική για το μέλλον. Το εάν τώρα είναι νομοθετημένη η εθελοντική είναι προφανώς μια απόφαση της ε, κάθε επικράτειας, αλλά η δουλειά του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικού ε, Κινδύνου σύμφωνα με την άποψή τους είναι πως ε, ο αποτελεσματικότερος μηχανισμό δημοσιότητας θα είναι ο ιδιωτικό τομέας με εθελοντική βάση και αν είναι μια βέλτιστη πρακτική θα υιοθετηθεί και από αυτού οι οποίοι εκδίδουν χρέο αλλά και αυτοί οι οποίοι παρέχουν κεφάλαιο θα το απαιτήσουν. Σας ευχαριστώ. Κύριε Σίχνμπουργκ, σας ευχαριστώ που ήρθατε. Στην ομιλία σας ε, το 2014 ε, είπατε πως ε, το 1931 επίσης το Ηνωμένο Βασίλειο είχε υψηλή ανεργία, ελλείμματα του προπολογισμού και χαμηλές αυξήσεις μισθών. Δεδομένου του ότι η Ευρώπη τα έχει όλα αυτά και περισσότερα ακόμα, το ότι αυξάνεται το εργατικό κόστος 5,9% σύμφωνα με τη Eurostat, ε, τα επίπεδα παραγωγικότητας πέφτουν, το εμπόριο ως ποσοστό του παγκοσμίου ΑΕΠ ε, πέφτει, ακόμα και στην καλύτερη χώρα στη Γερμανία έχουμε 7% ανεργία των νέων, στην Ελλάδα είναι πάνω από 50%, η μέση ανεργία είναι 11,6%. Όταν αναλύεται τους συστημικούς κινδύνους σε μια οικονομία στο σύνολό της, είτε είναι η Ευρωζώνη είτε είναι 28, λαμβάνεται υπόψη το ότι υπάρχει συστημικός κίνδυνος στο σκεπτικό και την οτροπία κάποιων ανθρώπων που εξετάζουν συνεχώς τις ίδιες λύσεις στα ίδια προβλήματα, την λεγόμενη περισσότερη Ευρώπη δηλαδή, αντί να σκεφτούν κάτι το εναλλακτικό. Και θα έλεγα επίσης το ότι όσον αφορά τις δυνατότητες εναλλακτική σκέψης, αντί να πάμε σε μια κεντσιανή φιλοσοφία που οδηγεί σε κορπορατισμό, μπορούμε να εξετάσουμε εναλλακτικά μοντέλα, είτε μιλάμε αν για ανεξάρτητες ε, χώρες και αν μπορούν να ανθίσουν πέρα από αυτή την νοοτροπία. Μια εναλλακτική πολιτική για τους ε, φόρους ε, ή την ανάπτυξη και τις δουλειές για να υποφεληθούν οι λαοί των χωρών αυτών. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση αυτή και για το ότι διαβάσετε μια ομιλία μου. Κοιτάξτε, όταν κάνω διάκριση μεταξύ χρόνιας και οξίας φάσης της ε, κρίσης, είχαμε την οξία φάση το 2010 μέχρι το 2012. Και πρέπει νομίζω να αναγνωρίσουμε από τη σκοπιά της ε, χρηματοπιστωτικής ε, σταθερότητας και του σχετικού κινδύνου όπως οφείλω να κάνω, πρέπει πρώτα απ' όλα να δούμε τους άμεσους κινδύνους που υπήρχαν και ήταν θα έλεγα υπαρξιακής φύσεως και έχουν συνέπειες για τις τράπεζες ε, και τις ε, χρηματαγορές και τα βήματα τα οποία κάναμε ε, από το 2010 μέχρι πρόσφατα και μείωσαν ε, κατά πολύ τον οξύ κίνδυνο χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και αυτό το είδαμε στα γεγονότα του Ιουνίου ότι υπήρχε μια κάποια προστασία και μόνωση του συστήματος λόγω της προόδου στην Τραπεζική Ένωση διαφόρων μηχανισμών προστασίας που υπήρχαν. Και άρα έχουμε το δεύτερο ερώτημά σας που αφορά θα έλεγα το, το χρόνιο ζήτημα δηλαδή τι προοπτικές υπάρχουν για να φύγουμε από την φάση αυτή της ανάρρωσης θα την χαρακτηρίζα. Θα έλεγα πως ε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου κοιτάει και την πρόοδο στις ε, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις οι οποίες είχαν αυξήσει κάπως ε, την αντοχή των οικονομιών της Ευρωζώνης ε, που εξορισμού είχαν μεγαλύτερη δυνατότητα απορρόφησης των σοκ. Οπότε αξιολογώντας τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές ε, δημοσιονομικής σταθερότητας ε, στην Ευρωζώνη πρέπει να γίνει μια αξιολόγηση και οπωσδήποτε η Τράπεζα της Αγγλίας, ε, το Συμβούλιο μας και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου αξιολογούν τις προοπτικές αυτές που είπαμε για την ανταγωνιστικότητα, το μισθολογικό κόστος κτλ. Οπότε υπάρχει αυτή η πρόοδος στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που οπωσδήποτε διαφέρει από χώρα σε χώρα και όπως αναφέρθηκε και η κύρια Φεράρα υπάρχει το ζήτημα και των λοιπών μέτρων που από μόνα τους θα βελτιώσουν την λειτουργία της Ευρωζώνης. Οπότε ναι πρέπει να ληφθούν αυτά υπόψη λέγοντας πως ε, σαφώς υπήρχε πρόοδος από τις χειρότερες στιγμές ε, της κρίσης μέχρι τη στιγμή που έβγαλε αυτόν τον λόγο και έκτοτε έχει υπάρξει και άλλη πρόοδος. Αλλά βεβαίως όπως παντού υπάρχει κάποιος κίνδυνος που παραμένει. Σας ευχαριστώ. Ε, Καλώς ήρθατε και ευχαριστούμε και για τις παρατηρήσεις ε, και για την παρουσίασή σας. Ε, θα ήθελα να σας κάνω διάφορες ερωτήσεις. Ε θα απαντήσετε με την ιδιότητα του πρώην πρόεδρου του SRB. Το είπατε στην προηγούμενη συνεδρία ότι υπάρχουν δύο βασικά ζητήματα για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Παραδείγματο χάρη δράση προτεραιότητα για τη φερεγγιότητα 2 και θα ήθελα να σα ακούσω σε σχέση με αυτό το θέμα. Όπως είπε και η κυρία Σουίνμπερν, όταν απαντήσατε είπατε ότι υπήρχαν κάποιες ανεπιθύμητες συνέπειες και δεδομένου του ότι χρειάστηκαν άπειρες νομοθετικές ρυθμίσεις ε, για να χειριστούμε το συστημικό κίνδυνο. Όταν εξετάζετε αυτά που έγιναν και βλέπετε την προσαρμογή των νομοθετικού χαρακτήρα αποφάσεων για να ε, ε, χειριστούμε το συστηματικό κίνδυνο, θεωρείτε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λειτουργεί καλά ως προς τις δυσλειτουργίες, κυρίως σε σχέση με το συστημικό κίνδυνο και τι πρέπει να γίνει στο μέλλον. Δεύτερον, ε, ξέρετε ε, τη κατάσταση στην Ιρλανδία, τη χώρα μου και το εύρος της κρίσης ε, στην αγορά των ε, κινήτων ήταν μια σημαντική παράμετρος που οδήγησε αυτή την ευρύτερη χρηματοπιστωτική κρίση. Ε, στη δουλειά που κάνατε στο Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου, όταν εξετάζατε τους κινδύνους στην αγορά κινήτων και από ό,τι κατάλαβα εξετάζετε τώρα τις βαθύτερες αιτήσεις και θα δημοσιεύσετε και ένα βιβλίο σε σχέση με αυτό. Ε, τι ε, πιστεύετε για τις ε, φορολογικές εκτόσεις, για, την, για, τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και πιστεύετε ότι υπάρχουν πιθανές συνέπειες και σε άλλες αγορές μπορεί να επέμβει τελικά η Ευρωπαϊκή Κεντρική η Τράπεζα για να παρεμποδίσει αυτές τις αρνητικές συνέπειες σε άλλους ε, τομείς της αγοράς. Απάντηση. Είπα ότι υπήρχαν κάποιες, κάποιες ανεπιθύμητες επιπτώσεις ε, του ΕΜΕΡ και των χρηματοπιστωτικών ε, κανονισμών και φαντάζομαι, όπως απάντησα και στην κυρία Σουίνμπερν, Όσο εξελίσσεται η κατάσταση και προσθέτονται νέα στοιχεία στο σύστημα, θα προκύπτει ε, διαρκώς η ανάγκη προσαρμογής. Ε, θα πρέπει να εξετάζουμε ε, διαρκώς την πορεία που διαγράφουμε από τον αρχικό σχεδιασμό μέχρι την νομοθεσία και τις, τους τομείς όπου που απέτυχε η νομοθετική ρύθμιση. Τι μπορεί να κάνει η ΕΚΤ, ρευστότητα και ευαλωτότητα των αγορών. Δηλαδή, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ε, παροδική ε, ε, έλλειψη ρευστότητας ε, και μετά ξαφνική αύξηση ρευστότητας. Γιατί συμβαίνει αυτό, υπάρχει ρυθμιστική αιτία ή απλώς αλλάζουν οι στρατηγικές θέσεις εμπορία ή συναλλαγών των βασικών φορέων των αγορών και ακόμη και σε άλλους θεσμούς, ε, το FSB, το ESB ε, και εκεί πέρα πέρα από την ΕΚΤΕ προσπαθούμε ακριβώς να πραγματευτούμε αυτό το ζήτημα και να διαπιστώσουμε αν ε, κατά τη γνώμη μας μπορεί να υπάρξει ένας λόγος μόχλευσης ή αλλαγές στη μήτρα ρευστότητας γιατί αλλάζει και η φύση των αγορών και έχουμε ένα συνδυασμό των darker pools και των ρευστών ε, των αγορών που λειτουργούν με ανοιχτή ρευστότητα. Ε, γίνεται μία έρευνα από πλευράς ε, του ESRB ε, για τις αγορές σε περίπτωση στρες, ενώ αντίθετα υπάρχουν 150 επενδυτικά ταμεία που διαχειρίζεται η Τράπεζα της Αγγλίας. Εμείς 2.000 θα ερευνήσουμε στα πλαίσια της μελέτης. Βλέπετε είναι διαφορετική η κλίμακα και έτσι θα φέρουμε νέα στοιχεία προς τη ρευστότητα των αγορών για τα σπίλοβες και τη ρευστότητα της αγοράς νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο να μιλήσω για αμοιβαιότητα. Τονίζεται η σημασία της αμοιβαιότητας. Δηλαδή, μια εθνική κεντρική τράπεζα, όπως αυτή της Ιρλανδίας παραδείγματος χάρη, να λαμβάνει μέτρα για να περιορίσει ε, τη ε, μήτρα της ρευστότητας σε σχέση με τα δάνεια στον τομέα των ακινήτων. Όμως, άλλες αρχές παίρνουν αντίστοιχα μέτρα και το παρακολουθεί ε, η ΕΚΤΕ και υπάρχει τότε ρυθμιστικό αρμπιτράζ. Ε, ξέρετε ότι από μέρα σε μέρα μπορεί να αλλάξει άρδινη κατάσταση και δεν ε, μπορούμε να έχουμε τέτοιο ρυθμιστικό αρμπιτράζ διότι για το αντικυκλικό buffer και για την αμοιβαιότητα έχουμε μηχανισμό, δηλαδή για ευρύτερα μακροληπτικά μέτρα έχουμε το κεντρικό clearing και γι' αυτό πρέπει να εξασφαλίζουμε ε, την ηρεμία στην αγορά και σας διαβεβαιώ όλοι θέλουμε να εξασφαλίζουμε την αρμονία και να αποφεύγουμε τα spillover σε άλλους τομείς. Ευχαριστούμε Νίνα Τζιλ. Ε, ευχαριστώ και καλωσορίσατε Τρία σύντομα σημεία θα ήθελα να σχολιάσω. Ε, μία σύντομη μελέτη δείχνει ότι ο τραπεζικός τομέας είναι στην εντατική ακόμη, διότι οι τράπεζες της Ευρωζώνης δεν σημειώνουν πρόοδο προς τον καθαρισμό, τον ισολογισμό τους ε, ένα χρόνο μετά τα τεστ εκοπόσεως. Λένε 886 ε, δις κόκκινων δανείων εξακολουθήσουν να υπάρχουν στους ισολογισμούς των τραπεζών της Ευρωζώνης και έχει επέλθει μείωση μόνο 2% τους τελευταίους 12 μήνες. Ε, το ESRB ε, ανησυχεί με όλα αυτά τα κόκκινα δάνεια και ε, τι πρέπει να κάνουν οι τράπεζες. Ταυτόχρονα τι κάνουμε ε, για να αποφύγουμε την τυπλοποίηση αυτών των ε, ε, ληξιπρόθεσμων δαμηνίων, διότι προσπαθεί να επαναφέρει την τυπλοποίηση η ΕΚΤ. Δεύτερον, τομέας ακινήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι ο τομέας μου, από εκεί έρχομαι και η κρίση των υπόθηκων δανείων δείχνει πόσο μη βιώσιμες είναι οι πολιτικές και πώς μπορούν να κλονίσουν ολόκληρη τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα. Πώ αποτιμάτε τις ε, συνέπειες, ε, πιθανές συνέπειες ε, της πολιτικής που προτείνει ο Υπουργός Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου για την σύναψη υψηλότερων ενυπόθηκων δανείων ώστε να αυξηθεί το ποσοστό της ιδιοκτησίας. Ιστορικά βλέπουμε ότι τα ενυπόθηκα δάνεια στο Ηνωμένο στη ΣΥΠΑ οδήγησαν σε καταστροφή και παρόλα αυτά συνεχίζεται η τιτλοποίησή τους ε, στη ΣΥΠΑ. Στο, το FSB ε, πρότεινε να μεταρρυθμιστεί η χρηματοοικονομική αγορά, ενέκρινε το, το Κοινοβούλιο το ψήφισμα του, το Συμβούλιο όμως ακόμη μετά από δυόμιση χρόνια συζητήσεων δεν μπορεί να καταλήξει η συμφωνία. Στο μεταξύ οι ΥΠΑ έχουν προχωρήσει. Ως πρόεδρος του FSB, σε ποιο βαθμό ανησυχείτε ότι είναι ουραγός η Ένωση ε, στα πλαίσια αυτής της παγκόσμιας ε, μεταρρύθμισης, ε, κυρίως ε, σε περίοδο χαμηλών επιτοκίων. Αυτά τα ταμεία θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν σταθερή αξία των υποκείμενων στοιχείων, διότι το είπατε ότι η Τράπεζα της Αγγλίας ασχολείται βεβαίως με τις δικές της σημαντικά, σημαντικές τράπεζες, αλλά εσείς ε, ελέγχετε 2.000 τράπεζες. Πολύ ωραία ερώτηση για, την, ε, τομέα, ε, για τον τομέα των τραπεζών. Κάθε φορά που συνεδριάζουμε στο ESRB ασχολούμαστε με αυτό το ζήτημα και Υπήρξε πρόοδος μετά από ε, την, ε, την αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού και τα ε, στρες, τα τεστ κοπόσεων που έγιναν για τις τράπεζες πριν από ένα χρόνο. Φυσικά για τις μεγαλύτερες τράπεζες χρειάζεται και πιο εντατική εποπτεία. Η ονομαστική αξία της ανάπτυξης είναι ιδιαίτερα χαμηλή στην Ευρώπη το τελευταίο χρόνο ε, και χρειάζονται κεφαλαιοποίηση οι τράπεζες ε, ως εκ τούτου και γι' αυτό κάναμε και την αξιολόγηση των ε, στοιχείων ενεργητικού και τα τεστ κοπόσεως. γενικό σχόλιο θα κάνω μόνο για το τραπεζικό τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ πιο υγιή στα τελευταία χρόνια. Δεν ε, έχουν αρθεί όλε οι ανησυχίε, αλλά είναι σαφώς υγιέστερος ο τομέας και βλέπουμε συγκεκριμένε συνέπειες. Ε, δηλαδή, υπάρχει ε, ανάπτυξη με θετικό πρόσημο τη δανειοδοσία και είναι σχετικά, παραμένει σχετικά φυσιολογική η ανάπτυξη, οπότε υπάρχουν απτά σημάδια βελτίωσης. Φυσικά επιδέχεται βελτιώσεις ε, ο τομέας. Για την ε, τιτλοποίηση και την αναδιάρθρωση, γιατί γι' αυτό πιστεύετε νομίζω, δηλαδή τα αναδιαρθρωμένα δεν να περάσουν σε διαφανείς τιτλοποίησεις, αυτό σχολιάσατε, νομίζω ότι αυτό ε, πρέπει να το προσέξουμε και εντάσσεται στα πλαίσια του STS. Το, η αγορά κινήτων Έχουμε αυτά τα προγράμματα Help to Buy, βοήθεια για αγορά σπιτιού. Είναι περιορισμένου εύρου σε σχέση με τον, το μέγεθος της αγοράς ακίνητων στο Ηνωμένο Βασίλειο και είναι καλά στοχευμένα, αποδεδειγμένα, βασίζονται σε, για, σε αγορά πρώτης κατοικίας και ε, επίσης κοιμούμαστε σε τιμές κάτω του μέσου όρου ε, και τα υποκείμενα ε, πρότυπα ε, επειδή έχουν γίνει και προσαρμογές ε, στα προγράμματα, αντιστοιχούν στο κίνδυνο που αναλαμβάνουμε, θεωρώ. Ε, στη, α, ναι, στην Τράπεζα της Αγγλίας, επειδή μας ζητάνε και αιτήσια αποτίμηση αυτών των προγραμμάτων, Δεν θα περιμέναμε την ετήσια επισκόπηση, ξέρετε, αν εντοπίζαμε ε, σοβαρή πηγή ανησυχίας, ε, αλλά σας λέω ότι σε σχέση με, το, σε σχέση με τα πρότυπα και την υποκείμενη αξία των υπόθηκων δανείων, δεν θα έλεγα ότι υπάρχουν ε, σημεία ανησυχίας και το Συμβούλιο σίγουρα έχει και τις προτεραιότητες του, γιατί έχει πολλαπλέ αρμοδιότητε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ και καλώς ήρθατε. Χαίρομαι και για το ότι βεβαίως ε, υπάρχει η δική σας εμπειρία στο Συμβούλιο αυτό και για το ότι ε, αφιερώνεται και χρόνο σε μας. Να αναφερθώ στο ερώτημα του κυρίου Λάμπερτς για το περιβαλλοντικό ζήτημα και τη φούσκα του άνθρακα γιατί ξέρετε πως αναφέρθηκε ο κίνδυνος ε, όσον αφορά την ε, τιμή που υπάρχει, τη δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα και οπωσδήποτε και η Τράπεζα της Αγγλίας έχει κοιτάξει τον τομέα των ασφαλιών. Βλέπω πως από την απάντησή σας δεν το θεωρείτε αυτή τη στιγμή ε, κέριο ζήτημα αλλά κάτι το μακροπρόθεσμο αλλά ταυτόχρονα λαμβάνονται αποφάσεις ειδικά αυτή τη στιγμή όσον αφορά την κατανομή επενδύσεων Οπότε θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό το ζήτημα. Πρώτα απ' όλα λοιπόν να σας ρωτήσω θεωρείτε πως ε, αυτή τη στιγμή υπάρχει κάποια αβεβαιότητα, κάποια πρόοδος ή όχι. Και ρωτάω τώρα καθώς το κόστος των ορυκτών καυσίμων είναι χαμηλό, το κόστος των εκπομπών επίσης, και έτσι μπορεί κάποιοι να λάβουν αποφάσεις ε, οι οποίες δεν θα είναι βιώσιμες ε, μακροπρόθεσμα. Δεύτερον, ορθώς αναφέρατε τον ρόλο των κυβερνήσεων και των ε, κοινοβουλίων. Αναρωτιέμαι λοιπόν εάν θεωρείτε πως οι κυβερνήσεις στέλνουν σωστά και ξεκάθαρα μηνύματα. Τέλος, στο Κοινοβούλιο ασχολούμαστε και θα συνεχίσουμε να ασχολούμαστε στο μέλλον με το σύστημα εμπορίας εκπομπών. Αναρωτιέμαι λοιπόν σε ποιο βαθμό η ορθή λειτουργία α, της ε, τιμής, ε, παραδείγματος χάρη, των ε, αδειών εκπομπών μπορεί να βοηθήσει την αγορά να αξιολογήσει σωστά τον κίνδυνο και να αποτιμήσει σωστά τα στοιχεία που υπάρχουν σε αυτό το τομέα. Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Όσον αφορά τον άμεσο κίνδυνο, δεν θα επαναλάβω την προηγούμενη απάντησή μου, κάπως ε, συγκεντρωμένο στον κλάδο των ασφαλιών. Αλλά υπάρχουν. Υπάρχει ένα στατιστικό στοιχείο, όπως ξέρετε, ότι ο αριθμός ακραίων καιρικών φαινομένων έχει αυξηθεί, έχει τριπλασιαστεί από το 1980. Οι ζημιές από αυτά τα φαινόμενα έχουν πενταπλασιαστεί, γύρω στα 5 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο, αποπληθωρισμένα πάντα. Οπότε μιλάμε για τάξεις μεγέθους. Ο κλάδος των ασφαλιών το είχε αντιμετωπίσει σωστά. Αλλά εκεί όπως είπα εκδηλώνεται το ζήτημα. Τώρα, αν, ε, ε, αν υπάρχει ευαισθητοποίηση για το ζήτημα, ναι, οπωσδήποτε. Και αυτή τη στιγμή βεβαίως πάει χέρι-χέρι με τις ανεπαρκείς ε, πληροφορίες για να διαχειριστούμε πλήρως το ζήτημα, αν είναι κάποιος π.χ. επενδυτής. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αν κάποιος έχει π.χ. ένα αρκετά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο να αποφύγει τον άνθρακα. Και αυτό το οποίο είναι δύσκολο ακριβώς είναι το να στοχεύσει σε εταιρείε οι οποίες έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα, κάτι το οποίο θα ήθελαν να κάνουν κάποιοι επενδυτές, αλλά δεν έχουν τις σχετικές πληροφορίες που φτάνουν στην ουσία του ζητήματος. Το θέμα τώρα για τα σαφή μηνύματα των κυβερνήσεων. Ε, εδώ έχουμε άλλο ένα πιθανό όφελος ε, της αυξημένης δημοσιότητας ε, στον ιδιωτικό τομέα, καθώς θα αποκαλύψει τον βαθμό στον οποίο οι εταιρείε έχουν μια στρατηγική για να μειώσουν το αποτύπωμα άνθρακα. Είτε αυτή η στρατηγική αφορά το εθνικό, τους εθνικούς στόχους ή κάποιον άλλο στόχο, αν δεν υπάρχει στρατηγική και αν δεν υπάρχει στρατηγική, κατόπιν μπορεί να είναι μια απόφαση, το εάν αυτό έχει συνέπειες μετά. αν ισχύουν όλα αυτά, δηλαδή δεν υπάρχει στρατηγική και δεν έχει αυτό συνέπειες όσον αφορά την πρόσβαση σε κεφάλαιο, σημαίνει πως υπάρχει μια έλλειψη αξιοπιστίας του συνολικού πλαισίου πολιτικής το οποίο πρέπει να λέει κάτι στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις για το αν απαιτείται κάποια περαιτέρω δράση. Βεβαίω ισχύει και το αντίστροφο ότι οι εταιρείε ε, με τις καλύτερες στρατηγικές θα αποτιμηθούν υψηλότερα και έτσι θα υπάρξει ένας και κύκλος κτλ. Τώρα, για λόγους χρόνου και εμπειρίας θα αφήσω εκτός το σύστημα εμπορίας εκπομπών. Ευχαριστώ. Γιάκοπ Φον Βάιστσέκερ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Διοικητά. Δύο ερωτήσεις. Η πρώτη αφορά την ενδιαφέρουσα ιδέα που αναφέρατε στην εισαγωγή του δυναμικού λόγου μόχλευσης. ξέρετε πώς διαβάζουμε τις ομιλίες σας. Σε μία από αυτές, ε, ως διοικητής της Τράπεζας Αγγλίας, είπατε πως εξετάσαμε το συνολικό επίπεδο κεφαλαίου. Θεωρούμε πως το σύστημα χρειάζεται είναι ακριβώς ε, το σύστημα θα έλεγα πως αντιμετωπίζει τις ανάγκες που υπάρχουν. Οπότε θα ήθελα να ακούσω από σας το εάν θεωρείτε πως κάποιες τέτοιες ε, διατάξεις για δυναμικό ποσοστό μόχλευσης θα μπορούσαν να βοηθήσουν και τι θα μπορούσε να υπάρξει σε ευρωπαϊκή νομοθεσία. Πρώτη ερώτηση είναι αυτή. Η δεύτερη είναι κάπως πιο πολιτική. Σχετίζεται με το TILAC. Έχω την αίσθηση, ειδικά στις Βρυξέλλες, πως κάποιοι ελπίζουν πως το ΤΙΛΑΚ θα μπορούσε να υποκαταστήσει το ΕΜΡΕΛ και διάφορα άλλα νομοθετήματα. Δεν ξέρω λοιπόν πως το ΤΙΛΑΚ μπορεί να συμπληρώσει τα άλλα δύο νομοθετήματα αντί να τα υποκαταστήσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάλιστα. Μπήκατε στην ουσία του πρώτου θέματος ε, στην απόφαση της Επιτροπής ε, Δημοσιονομικής Πολιτικής ε, της Τράπεζας Αγγλίας θεωρήσαμε πως το σύστημα είναι επαρκώς κεφαλαιοποιημένο ή να είναι πολύ κοντά στο στόχο αυτόν μιλάμε για λιγότερο από 1% όπως είχαμε πει τότε Τώρα για κάποιους λόγους. Πρώτον κοιτάξαμε την εμπειρία των προηγούμενων ε, χρηματοπιστωτικών κρίσεων ε, όπως έγινε βεβαίως και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Βασιλεία και αλλού. Αλλά δεύτερον βασιζόμαστε σε δύο στοιχεία που θα είναι μέρη του συστήματος. Το πρώτο είναι αξιόπιστη TILAC και EMREL. Δηλαδή τη δυνατότητα απορρόφησης ε, ζημιών η οποία βεβαίως οδηγεί σε κάποια πειθαρχία αλλά οδηγεί και σε πιο αποτελεσματικές κεφαλαιακές δομές και το δεύτερο είναι η ενεργή χρήση του αντικυκλικού αποθεματικού και για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί με το αποθεματικό αυτό εμείς θεωρούσαμε πως χρειάζεται ένα υψηλότερο, ένας υψηλότερος λόγος μόχλευσης. Και βεβαίως χρειάζεται μια πιο συνεκτική και αποτελεσματική και δομή. Γιατί αν δεν υπήρχε αυτό θα χρειαζόταν να σωρεύουμε συνεχώς επιπρόσθετο κεφάλαιο και με τον ίδιο τρόπο θα αντιμετωπίζαμε και την μη μόχλευση κτλ. Το θέμα λοιπόν του δυναμικού λόγου μόχλευσης που αγούγεται κάπως περίπλοκο κατά βάση είναι να διασφαλίσουμε πως τα κίνητρα αυτά αυξάνονται με τη σειρά τους εάν αυξάνεται και το αποθεματικό. Να σας δώσω το παράδειγμα του Ηνωμένου Βασιλείου. Το τυποποιημένο μοντέλο, μοντέλο για κινδύνου για τα ενυπόθηκα δάνεια είναι 35%. Το αντίστροφο αυτού είναι επί 3. Όταν προσθέτουμε κεφάλαιο, επειδή μια τράπεζα είναι συστημική ή για άλλους λόγους, αυξάνουμε το ποσό κεφαλαίου σύμφωνα με μια στάθμιση κινδύνου. Εάν το, η στάθμιση παραμείνει η ίδια, σημαίνει πως ε, κινδυνεύουμε περισσότερο. Εάν λοιπόν αυξήσουμε και τα δύο ταυτόχρονα, κατά 35 μονάδες ε, βάσης, ε, όπως είπα, τότε παραμένει σταθερή η αναλογία. Αυτό είναι ουσιαστικά το, το νόημα εν ολίγης. Όσον αφορά τώρα την τελευταία σας ε, ερώτηση, θα απαντούσα ως εξής ειδικά σε σχέση με το BRD και τα στοιχεία του νομοστήματος αυτού. Το κεφάλαιο από μόνο του και η δυνατότητα απορρόφησης ζημιών είναι αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη για να μην υπάρχουν τραπεζικά ιδρύματα που είναι πάρα πολύ μεγάλα για να χρεοκοπήσουν. Ειδικά για τα πάρα πολύ μεγάλα απαιτούνται διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Πρέπει να υπάρξει τρόπος σε μια διάσωση ή λύση αυτών των τραπεζών ε, μια απομόνωση των βασικών λειτουργιών τους ε, και βεβαίως δεν υπάρχουν διαφορετικές δομές σε διαφορετικές χώρες. Για να τελειώσω λοιπόν, στο επίπεδο του δικού μας του Συμβουλίου για οποιοδήποτε συστημικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που έχουν έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση περνάνε αυτή τη διαδικασία αξιολόγησης, όπως λέγεται, της διαδικασίας διασώσης, όπου κοιτάμε όχι μόνο το ποσό του κεφαλαίου έχουν, αλλά πού το έχουν, τι λακ κτλ έτσι ώστε να υπάρχει μια αξιοπιστία σε μια διαδικασία όπως είπαμε διάσωσης για να είναι αξιόπιστη η διαδικασία σε επίπεδο εγχώριο και παγκόσμιο. Σίγκφριντ Μουρεσάν. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, καταρχήν ε, για την αγορά ακινήτων. Νομίζω το Σεπτέμβριο στο Γενικό Δικτικό Συμβούλιο της ΣΕΚΤ είπατε ότι σε σχέση με την αγορά κινήτων χρειαζόταν περισσότερη εργασία και θα έπρεπε να γίνει αυτό από την ΕΣΡΠ στους επόμενους μήνες και τα αποτελέσματα θα δημοσιεύονταν. Υπήρξαν λοιπόν, υπάρχουν μάλλον εξελίξεις που παρατηρείται στην αγορά κινήτων της Ευρώπης, ιδιαίτερα υπό το φως των χαμηλών επιτεκίων για τα ενυπόθηκα δάνεια και την έλλειψη δράσης στα εμπορικά ακίνητα. Και μήπως από τις εργασίες που κάνετε μπορείτε να μας διαφωτίσετε. Δεύτερον, για την ποσοτική χαλάρωση που συνδέεται με τις μακροπροληπτικές απαιτήσεις αυτό έγινε για να ενθαρρυνθεί ο δανεισμός και να αντισταθμιστούν τα χαμηλά επιτόκια. Όμως οι συνάδελφοι λένε ότι οι μακροπροληπτικές απαιτήσει στην ουσία υπονομεύουν την ποσοτική χαλάρωση στην Ευρώπη. Ποια είναι η δική σας άποψη γι' αυτό και πόσο καλά λειτουργούν από κοινού αυτά τα δύο μέσα και συνδυασμένα οδηγούν στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Τέλος, στην τελευταία διάλογο με τον Μάριο Ντράγκη μας είπε ότι υπήρχε ένα ικανοποιητικό επίπεδο στο οποίο θέσπιζαν ε, το πλαίσιο μακροπροληπτικής ε, εποπτείας ε, τα κράτη-μέλη, εκτός από την Ρουμανία, και την Ιταλία και το Βέλγιο. Και μάλιστα μας είπε ότι πιέζει τις χώρες αυτές για να ενημερώσουν την νομική, τη σχετική νομική βάση. Υπάρχουν νέα γι' αυτό. Ευχαριστώ. Όσον αφορά την αναθεώρηση των μακροπροληπτικών προβλέψεων για την αγορά ακινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε ότι υπάρχουν διαφορές στις αγορές αυτές. Σε κάποιες αγορές οι αρχές ήδη έχουν προβεί σε δράσεις μακροπροληπτικές. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μία από αυτές. Η Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής προέβησε δράση ώστε να δοθούν δάνεια στα νοικοκυριά Επίσης εισήχθη, εισήχθηκαν μάλλον έλεγχοι δοκιμές για ε, δάνεια χαμηλού επιτοκίου. Έχουν γίνει και άλλες δράσεις όπως ας πούμε κάποιες φορολογικές αλλαγές που αντίθετα με την προηγούμενη συζήτηση που αφορούσε συγκεκριμένα προγράμματα ώστε να δοθούν κίνητρα στους νέους αγοραστές αυτές οι φορολογικές αλλαγές αναμένεται να ε, οθήσουν τις δραστηριότητες σε κάποιες πτυχές της αγοράς. Με την Τράπεζα της Αγγλίας, το PRA, κάνει μία ε, έρευνα όσον αφορά την αγορά των ε, ιδιοκτητών ώστε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξει πτώση των τιμών. Ε, για την ώρα δεν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις. Πάντως το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ένα παράδειγμα δικαιοδοσίας όπου έχουν ληφθεί μέτρα, έχουν ε, αποφασιστεί πράγματα και είναι χρήσιμο η SRB να κάνει μια ευρύτερη μελέτη, ευρύτερη επισκόπηση ώστε να υπάρχουν σχετικά σχόλια τους επόμενους μήνες. Για τα εμπορικά ακίνητα, οι αξιολογήσεις έχουν κυμανθεί σε μεγάλο βαθμό σε διάφορες δικαιοδοσίες. Να μιλήσω για το Ηνωμένο Βασίλειο ότι ο βαθμός μόχλευσης στο σύστημα και των ε, χρηματοπιστωτικών, ε, των βρετανικών χρηματοπιστωτικών ε, ιδρυμάτων δεν έχουν μεταβληθεί. Δηλαδή, με άλλα λόγια, έχουν έρθει, έχει έρθει ξένο χρήμα στην αγορά. Παρακολουθούμε δε και τις εξελίξεις ε, ε, όσον αφορά την αγορά, τις αγορές των ε, ομίλων ή καταπιστευμάτων για τα ακίνητα και δεν προβαίνουμε σε κάποιες συγκεκριμένες ενέργειες. Από την πλευρά βέβαια της SRP όντως πρέπει να παρακολουθείτε η κατάσταση. Τώρα, συμβατική νομισματική πολιτική και η σχέση αυτής με την μακροπροληπτική πολιτική. Εν γέννη, η μακροπροληπτική πολιτική, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων, μπορεί να είναι παραπληρωματική ώστε να κινητοποιήσει την νομισματική πολιτική. Δηλαδή, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν σε αγορές ακινήτων, όπως είπατε πριν από λίγο, ενώ ταυτόχρονα προσπαθούμε να επιτύχουμε το στόχο ε, πληθωρισμού. Στην περίπτωση της ΕΚΤ είναι 2%. στην περίπτωση της Τράπεζας της Αγγλίας 2% ε, σε σχέση με τον πληθωρισμό. Ε, αυτό κάνουμε, δηλαδή η νομισματική αρχή ακατανοεί τι κάνει η μακροπροληπτική αρχή, ώστε να μπορούμε να σταθμίσουμε τις πολιτικές αναλόγως. Θα υπάρξουν περιπτώσεις, τώρα δεν, είναι, δεν ισχύει κάτι τέτοιο, όπου η νομισματική πολιτική και η μακροπροληπτική πολιτική μπορεί να λειτουργούν η ε, μία σε αντίθεση την άλλη. Αυτό δεν συμβαίνει όμως αυτή τη στιγμή. Όσον αφορά τις ενημερώσεις, και το νομικό πλαίσιο για τη μακροπροληπτική ε, πολιτική. Έχουμε αργότερα το, αυτό το μήνα συνάντηση με την SRB ε, και βεβαίως οι εν λόγω χώρες θα σχολιάσουν σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που προβλέπουν. Ευχαριστώ. Η αναλύση τότε. Ευχαριστώ. Αναφερθήκαμε σε διάφορες από τις ομιλίες σας σήμερα. Από τις μου πρέπει να πω ήταν οι, οι, ε, οι ομιλίες σας στο θέατρο Σέλντον είναι και στην πόλη μου, αλλά αυτό όχι μόνο επειδή ωραία μιλήσατε εκεί, αλλά και επειδή μιλήσατε για τις υποθέσεις της περιοχής μας, αν και προσέξατε να μην μπείτε στην πολιτική. Εμείς θέλουμε να αναπτύξουμε προληπτική κομμηχανισμό, όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να το κάνει αυτό μετά από την, ε, μεγάλη, μετά από την ύφεση την μεγάλη. Ε, όπως θα γνωρίζετε, υπάρχει αρκετή επίκριση σε σχέση με τις απόπειρες να δημιουργηθεί διαχωρισμός των τραπεζών, των, ε, των δραστηριοτήτων των τραπεζών για να προστατευτεί ο καταναλωτής. Αυτός που έχουμε δει όμως είναι ότι επηρεάζονται οι επενδύσεις. Ποια είναι η δική σας αξιολόγηση, ιδιαίτερα σε σχέση με αυτές τις ε, απόπειρες ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για διαχωρισμό των ε, δραστηριοτήτων των τραπεζών. Βλέπετε να είναι επιτυχής. Και επί το κύριο Νίδερ Μάγερ και ο κύριος Λάμπερτς απαντήσατε τις ερωτήσεις τους από την προπτική του FSP και εσείς ηγείστε το συζητήσεων ε, για τα αξιόγραφα, ε, ε, για τα κίνητα, με Αλλά από την SRB μήπως θα ήταν λογικό να υποστηρίξουμε πιο δεσμευτικά και τις προδιαγραφές, καθώς έχουμε ευρωπαϊκούς μηχανισμούς ώστε να τηρούνται οι περιβαλλοντικές προδιαγραφές που ισχύουν. Τώρα, όσον αφορά τα μπόνους των τραπεζιτών και δεν θα αναφερθεί σε αυτό τώρα, πάντως το πλαίσιο είναι ότι, δεν πρόκειται μόνο με τα μπόνους τα οποία συνδέονται με το κίνδυνο και την ανταμοιβή. Όσοι αναλαμβάνουν ευθύνες σε σχέση με τις πληρωμές θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούν μέσα στην οδηγία για τους ε, μετόχους πρέπει να κάνουμε περισσότερα έτσι ώστε οι χώρες οι οποίες δεν έχουν τέτοιου είδους ε, καθεστώτα να μην χρειάζεται να αναλάβουν την ευθύνη των ίδιων των μετόχων. Ναι. Μάλιστα, θα προσπαθήσω να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Για τη δεύτερη σας ερώτηση να προσπαθήσω να απαντήσω πρώτα, γιατί θεωρώ πως είναι περισσότερο θέμα διαδικασίας Νομίζω πως το ανέφερα και στις παρατηρήσεις μου στις εισαγωγικές. Η ESRB θα ασχοληθεί με αυτό το θέμα στο πρόγραμμα εργασίας του 2016, δηλαδή τους κινδύνους μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλού λύση κατανάλωση άνθρακα. Είμαι βέβαιο ότι ο πρόεδρο Τράγκη θα είναι πολύ πιο άνετο όταν θα έχει αυτή την ανάλυση και όταν θα έχει περισσότερη προοπτική για το θέμα. Είναι πάντως προτεραιότητα και σίγουρα θα εξεταστεί εις βάθος. Τώρα, όσον αφορά τις αμοιβέ των ε, τραπεζιτών, Εγώ έχω κάπως διαφορετική προοπτική και άποψη και νομίζω πως η προοπτική δεν είναι σημαντική γιατί αυτό που ήταν παλιά ένα μπόνους, δηλαδή πληρωμή σε μετρητά σε ένα συγκεκριμένο άτομο για μια χρονιά εργασία που του δινόταν στο τέλος του έτους και έπειτα ε, ήταν δικό του αυτά τα χρήματα ό,τι και αν ήταν αυτά τα μπόνους, ακόμα και αν είχαν ας πούμε, πληρωθεί μια προκαταβολή επί ενός συγκεκριμένου κινδύνου, μπορεί κάποιο τρόπο να είχαν για να πληρώσουν για αυτά τα χρήματα. Πάντως ε, ε, το, η κατάληξη είναι στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ότι ένα μπόνους που είναι η ανταμοιβή για, μιας, ε, για, για ενός χρόνου δουλειά, ένα κομμάτι αυτού, ένα, μια αναλογία αυτού ε, παρακρατείται ανάλογα με το... Μάλλον, και μετά επαληθεύεται κατά πόσο αυτό συνδέεται με την ανάληψη κάποιου κινδύνου ή όχι. Έτσι ώστε να προωθηθεί η μη επικίνδυνη ε, δραστηριότητα. Δηλαδή εξακολουθεί να υπάρχει ένα μπόνους, αλλά όχι με την έννοια που ισχύει το 1900, τη δεκαετία του 80. Προσπαθούμε λοιπόν να το διαχειριστούμε με τη λογική ότι αν μπορούσαμε περισσότερα να κρατήσουμε από την αμοιβή τους ετησίως, θα τους δώσουμε κίνητρα για να κάνουν το σωστό, να ενεργήσουν σωστά. Και αυτό που είδαμε με βάση τα στοιχεία που έχουμε από τότε που άρχισε να ισχύει αυτή η νομοθεσία είναι ότι η αμοιβή είναι η ίδια και ελαφρώς έχει αυξηθεί, αλλά το ποσοστό αυτό που μπορούμε να παρακρατήσουμε αν κάποιος έχει αναλάβει υπερβολικά πολύ κίνδυνο είναι μεγαλύτερο. Τώρα για την προστασία, την περιχαράκωση, το ring fencing και το πόσο αποτελεσματική είναι. Νομίζω πως η προσέγγιση που έχουμε είναι να φτιάξουμε ένα φραγμό, ένα ε, περιορισμό ανάλογα με το αν είναι κανείς ε, στο Λονδίνο, στη Γλασκόβη, αν είναι επιγραμμικά ή στο ε, εμπορικό δρόμο προς το συγκεκριμένο άτομο, στη λιανική πώληση, να είναι απόλυτα προστατευμένο να έχει ψηλότερη κεφαλαιοποίηση, όπως γνωρίζετε, από ότι το υπόλοιπο τραπεζικό σύστημα έχει συγκεκριμένη ευθύνη για την τράπεζα ε, προστασίας, ας πούμε, που προστατεύει και εμείς τους καλύπτουμε γιατί εξασφαλίζουμε ότι αυτή η πρώτη τράπεζα προστασίας, ό,τι και αν γίνει στην αγορά, το συγκεκριμένο ε, τραπεζικό ίδρυμα θα συνεχίσει να λειτουργεί και το Σαββατοκύριακο και στις επόμενες μέρες και χρόνια κτλ. Και Διστάζω τώρα να το συγκρίνω με μια συζήτηση που βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο και που μόνο θα ενισχύσει αυτό το σχόλιο ότι δηλαδή αυτό που είπε και ο κύριος Βαϊτζακέρ προηγουμένως ότι δηλαδή ότι το κεφάλαιο δεν αρκεί ώστε να υπάρχει και η ε, φερεγγιότητα και η ρευστότητα, αλλά θα πρέπει να συνδέεται με τη δυνατότητα εξυγίανσης και διάσωσης. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και για τα σχόλιά σας που είναι εξαιρετικά χρήσιμα για την εργασία μας εδώ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό και προσβλέπουμε στη συνέχιση της ε, ε, ανταλλαγής απόψεων μαζί σας όσο ε, γίνεται περισσότερο. Ευχαριστώ. Very well, dear colleagues. Let's move to point four of the agenda. πάμε στο σημείο 4 της ημερήσιας ε, διάταξης. Ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Βάλτερ Ράντερμάχερ, Γενικό Διευθυντή της Eurostat. Ευχαριστούμε που ήρθατε και χαιρόμαστε που ξεκινάει έτσι ο επίσημος ε, διάλογος για ζητήματα στατιστικής μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Eurostat, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για να δούμε ακριβώς ε, ποια θα είναι η υποπτία των δραστηριοτήτων αυτών της Κομισιόν, για να έχουμε αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία. Έχουμε και νομοθετικό διάλογο. Ο ένας βασικά έχει ολοκληρωθεί και υπάρχει ένα σημείο που εκρεμεί, που ελπίζουμε ότι μπορεί να επιληθεί. Και ένας άλλος έχει ξεκινήσει και όπως ξέρετε έχει μπλοκάρισε στο άλλο κομμάτι στο συνομοθέτη αλλά γενικά χαιρόμαστε για αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Θα δώσω λοιπόν τον λόγο στον κύριο Ραντερμάχερ και μετά θα ακούσουμε ερωτήσεις και απαντήσεις. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, μεγάλη μου τιμή που είμαι εδώ σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντικό για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Στατιστικών. Επίσημα εγκαινιάζουμε σήμερα τον επίσημο τακτικό διάλογο για τα στατιστικά ζητήματα και πριν από ένα χρόνο έγινε ο τριμερής διάλογος ε, για αυτό. Έγινε πέρυσι λοιπόν ε, του Αγίου Νικολάου το, ε, ο τριμερής διάλογος και πάλι ακριβώς ένα χρόνο μετά και μία μέρα ε, αρχίζει ο τακτικός διάλογος. Φοβερή πρόοδος. Ε, και είναι σημαντικό το ζήτημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Θα θυμάστε τις εντατικότατες διαπραγματεύσεις που μας οδήγησαν σε αυτό το σημείο. Δύο-τρία χρόνια χρειαστήκαμε. Κυρίως εσείς ε, κύριε Γκουαλκέρη και κύριε Μπαγιέ δεν τον βλέπω εδώ όμως. που είχαν σημαντική ε, συνεισφορά, ώστε να ε, ε, περατωθούν με επιτυχία αυτές οι δύσκολες μεν, αλλά τόσο σημαντικές διαπραγματεύσεις για τη στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή. Ε, ο κανονισμός του 2003 που άρχισε να ισχύει φέτος το Μάιο είναι η έκφανση της πραγματικής αλλαγής στην διακυβέρνηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα στατιστικά στοιχεία. Υψηλή ποιότητα, λογοδοσία, διαφάνεια. Αυτός είναι ο γενικός κανόνας για όλες τις στατιστικές αρχές. Ε, με αυτή την αναθεώρηση του κανονισμού ε, Το κανονισμό 2003, την ενιαία πράξη δηλαδή, θεσπίζουμε ένα σύστημα χάρη στο οποίο εφαρμόζεται πλήρως το άρθρο 338 των Συνθήκων Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι χάρη σε αυτό το σύστημα έχουμε το βέλτιστο δυνατό συντονισμό και βέλιστη δυνατή συνεργασία ανάμεσα στις στατιστικές αρχές τόσο εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτή η ενισχυμένη διακυβέρνηση οδηγεί ε, σε νέο ρόλο της Eurostat και του Διευθυντή της. Ε, είμαστε επικεφαλής του Ευρωπαϊκού ε, Συστήματο Στατιστικών Στοιχείων ε, και ε, ε, έχουμε ως πολιτικό συνομιλητή την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να τονίσω ότι αυτή η νέα αρχιτεκτονική είναι ιδιαίτερα ισχυρή ακριβώς επειδή είναι απλή και επειδή κατανοούμε σωστά οι ρόλοι. Έτσι κατοχυρώνεται η αποτελεσματικότητα διαφανή και λογοδοσία του συστήματος στις οποίες όλοι αποσκοπούμε. Αυτό το πρωτοποριακό ε, σύστημα θα πρέπει πλέον να εφαρμοστεί στην ε, πράξη και σε όλους τους τομείς. Ε, θα χρειαστεί να προσαρμοστούν στη νέα αρχιτεκτονική οι δομές που χρησιμοποιούν όλες τις στατιστικές αρχές. Από τότε που ήρθα και μίλησα για αυτό το θέμα το 2013 έχουμε αναλάβει διάφορες πρωτοβουλίες για να ενισχύσουμε την ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας και βλέπουμε ότι έχουν αποφασίσει φέρει σε οι προσπάθειές μας. Ε, θα ήθελα να σχολιάσω τρία ζητήματα συγκεκριμένα. Πρώτον, το επεισόδιο της Ελλάδας του 2009. Αυτό ήταν το δεύτερο βέβαια οδήγησε σε σοβαρά προβλήματα ε, φήμης και αξιοπιστίας των στατιστικών μας συστημάτων επαναλαμβανόμενο πρόβλημα σε μια χώρα η οποία, το οποίο πέρασε τα σύνορα και έπληξε την αξιοπιστία των ευρωπαϊκών στατιστικών στοιχείων για ολόκληρο το ευρωπαϊκό στατιστικό σύστημα. Spillover, παράπλευρη επίπτωση η οποία οφείλεται στην Ολένα και αυξανόμενη ολοκλήρωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από το 10 και μετά έγιναν νομικές μεταρρυθμίσεις και παρασχέθηκε τεχνική υποστήριξη προς την ΕΛΣΑ, την Ελληνική Στατιστική Αρχή, χάρη στο οποίο μπόρεσε να, να βαθμιστεί η ποιότητα των στατιστικών στοιχείων της, Ευρωπαϊκής Ελλάδας, πλέον ε, δεν υπάρχουν από το 2010 και μετά αμφιβολίες για τα στοιχεία που δίνει η ε, Ελλάδα. Ε, φυσικά χρειάζονται πολιτικές ε, αποφάσεις για να ε, επικυρωθούν τα θετικά αυτά αποτελέσματα. Ο διορισμός του νέου διευθυντή της Ελστάτε και η αναθεωρημένη νομοθεσία για την εκπόνηση στατιστικών στοιχείων συγκεκριμένα. Όμως ο, αδίκως υπάρχει μια επιθετικότητα σε επίπεδο εσωτερικού διαλόγου και αυτό εμποδίζει την ανάκτηση της αξιοπιστίας στο ελληνικό στατιστικό σύστημα και την αναγνώριση της μέχρι τούδε πρόοδου. Ε, θα πρέπει λοιπόν να ε, καταβάλουμε προσπάθειες σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη και η διαφάνεια και η λογοδοσία πρέπει να είναι βασικές αρχές. Ε, το 2011 με την δέσμη των έξι οδηγιών ε, δόθηκαν τα εργαλεία για ε, αυστηρή παρακολούθηση του υπερβολικού ελλείμματος σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, αυτό συνοδεύεται με αρμοδιότητες για την επιβολή των κυρώσεων και η νέα εντολή και οι νέες αρμοδιότητες θα ασκηθούν με ιδιαίτερη προσοχή και αιτιολόγηση ως προς την διαφάνεια που απαιτείται και την αναλογικότητα των μέτρων σε, σχέση, σε περίπτωση γνώμη επαναλαμβανόμενων υπερβολικών ελλημάτων. Ε, ε, είδαμε ε, στα στοιχεία του συστήματος υγείας από τη Βαλένθια, από την Ισπανία, κάποιες δυσλειτουργίες, κάποια πλημελή στοιχεία, τα οποία όμως ήταν περιορισμένα αλλά και επαναλαμβανόμενα δυστυχώς. Στενή συνεργασία με την Ισπανική Αμερικανική Στατιστική Αρχή μας βοήθησε να διορθώσουμε και να ανατάξουμε το σύστημα. Ήταν πολύ περιορισμένα αυτά τα επεισόδια και στο Συμβούλιο υποδεχτήκανε με ιδιαίτερη ικανοποίηση την συνεργασία ε, που προσέφερε η Ισπανική Αρχή. Αυτά εντάσσονται την ε, πολιτική εντολή που έχει δοθεί. Υπάρχει λοιπόν αποδοχή αυτής τη εντολής. Ε, τρίτον, συνεχίζουμε την στρατηγική μας ε, για τον εξυγχρονισμό του νομικού, τη νομική δομής ε, του ελληνικού στατιστικού συστήματος. Προσπαθούμε να επιτύχουμε πηγές σε συνδυασμό των πηγών, των δεδομένων τους, ώστε να αποφεύγουμε τις επικαλύψεις και να παραμένουμε ευέλικτοι. Υπάρχουν ε, διάφορες προτάσεις που θα κατατεθούν του χρόνου και στόχο θα έχουν να εξυγχρονίσουν και πάλι τη νομική δεδομή ε, ε, στο τομεί των επιχειρήσεων, της γεωργίας και των κοινωνικών αρχών. Το πρόγραμμα Levit για το οποίο έχουν αναλάβει σοβαρή δέσμευση και το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι κάτι που θα προωθήσουμε το 2016. Επίσης ανακοινώσαμε ε, τη, μία στρατηγική για την εκπόνηση των ευρωπαϊκών στοιχείων παρουσιάζοντας ε, το όραμά μας για τα επόμενα χρόνια έχει ε, εξελιχθεί αυτό το όραμα στο όραμα μέχρι το 2020 που ονομάζεται ESS, Ευρωπαϊκά Στατιστικά Στοιχεία, ε, ε, με διαφορετικές μεθόδους εκπόνησης στοιχείων και συλλογή στοιχείων, μια αλλαγή συστημικής σημασίας, αμοιβαίως επωφελής για όλους τους συμβαλόμενους φορείς, οι οποίοι θα ε, μπορέσουν να αντισταθμίσουν έτσι την έλλειψη πόρων από την οποία πλήττονται. Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Σα Σας είπα ότι η αποτελεσματικότητα και η πρόοδος είναι συνάρτηση της πολιτικής υποστήριξης και της σωστής εφαρμογής. Πρόσφατα κληθήκατε να συμφωνήσετε για πολύ σημαντικά ζητήματα, όπως είπε ο πρόεδρος παραδείγματος χάρη, η αναθεώρηση του ε, ο τιμών καταναλωτή ε, και υπάρχει και μία νέα πρόταση για ε, ε, πλαίσιο ποιότητα των στατιστικών στοιχείων σε σχέση με τη διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών. Επίσης, η έκθεση ΠΟΠ καλύπτει δύο βασικούς τομείς για την εκπόνηση πολιτικών για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων και δεν χρειάζεται όμως συνολική μεταρρύθμιση κατά τη γνώμη μας, διότι δεν, ε, ε, από τεχνικής πλευράς δεν έχει οριμάσει η πρόταση. Θα πρέπει να διευκολύνουμε απλώς ε, την εφαρμογή με απλωστευμένη διακυβέρνηση βάσει και του κανονισμού 223 και χρησιμοποιώντας τα όργανα της δευτερογενούς νομοθεσίας πέρα από τις συνθήκες. Συνεχίζονται διαπραγματεύσει. και είμαι πεπισμένος που μπορούμε να καταλήξουμε σε ικανοποιητικές συνενετικές λύσεις και για τον Πόπ και για το EHCP. Ε, η πρόταση για τα ΜΥΠΣ για τις μακρονομικές ανισορροπίε είναι πιο φιλόδοξη. Θα πρέπει να είμαστε ρηξικέλευθοι και με να καταφέρουμε να έχουμε ένα ενιαίο πρότυπο εξασφάλιση της ποιότητα για τα στοιχεία που αυτή τη στιγμή συλλέγουν τα, οι εθνικές στατιστικές αρχέ και να τα συνδυάζουμε με αυτά ε, που συλλέγουν σε κάποια κράτη-μέλη οι κεντρικέ τράπεζε, Γι' αυτό και είναι τόσο περίπλοξη διαπραγματεύσεις ε, και δεν με εκπλήσει το ότι υπάρχει στεναρή αντίσταση στο Συμβούλιο. προ το παρόν οι διαπραγματεύσει δεν έχουν οδηγήσει σχεδόν σε καθόλου πρόοδο. Ε, ποιος είναι ο στόχο μα να έχουμε εξασφάλιση τη διαφάνειας και τη λογοδοσία ε, για όλους τους δείκτες ε, μακροοικονομικών ισορροπιών για το ευρωπαϊκό σκορπό, τον πίνακα βαθμολογία, ανεξαρτήτω από τι αρχές, που εκπονεί τα στατιστικά στοιχεία δεν μπορέσουμε να συμφωνήσουμε τα πρότυπα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί αυτό ε, σχετίζεται και με τα δεδομένα που συλλέγουν ευρωπαϊκέ κεντρικέ ε, τράπεζες, τότε θα υπάρξει ένα κενό ω προ την διαφάνεια και τη λογοδοσία. αυτό, το, το εύρος αυτού του κενού, αυτού του χάσματο θα πρέπει να καλυφθεί από τα κράτη-μέλη και σύν χρόνο θα εξαρτηθεί η επιτυχία από τι εθνικέ ε, αποφάσει που θα ληφθούν βάσει αρχής επικουρικότητας. Σε ποιον θα αποδοθεί λοιπόν η ευθύνη για την εκπόνηση δεδομένων που θα σχετίζονται με τι μακροοικονομικές ανισορροπίε. Γι' αυτό σα λέω ότι χρειάζεται η ισορροπία ανάμεσα στους εξή παραμέτρους. Πρώτον, διαφάνεια και ποιότητα ε, των δεδομένων που παραγόνται σε σχέση και με τη διαδικασία εντοπισμού μακροοικονομικών ανισορροπιών και ε, μεγάλου ελλείμματο. Δεύτερον, στοιχεία που ε, πρέπει να παράσχουν τα συμβαλόμενα μέρη, άρα οι κεντρικέ τράπεζε και και τρίτον, τα στοιχεία που παρέχουν οι εθνικές αρχές. Ε, χρειαζόμαστε ισορροπία ανάμεσα στι τρεις παραμέτρους για να έχουμε την ε, ευκτία διαφάνεια, κυρίως, ε, ξαναλέω, για τι μακροοικονομικές ανισορροπίες. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να υποστηρίξουμε το θεσμικό ρόλο αυτής της διαδικασίας. Θα ήθελα τώρα, κλείνοντα. Να σας θυμίσω ότι στην πρώτη ανεπίσημη ανταλλαγή επόψεων με την Επιτροπή ΕΚΟΝ ε, μπόρεσα ήδη να σε ευαισθητοποιήσω για το πόσο ε, ραγδαίες ε, και σημαντικές είναι οι εξελίξεις που σημειώνονται όσο προσπαθούν να προσαρμοστούν στη νέα κατάσταση οι εθνικές στατιστικές αρχές. Το τωρινό σύστημα εκπόνηση στοιχείων πρέπει να προσαρμοστεί για να μπορέσει να ανταποκριθεί στην εντολή που δίνεται. Χρειάζονται μεγαλύτερες, περισσότερα και καλύτερα δεδομένα ε, και χρειάζεται καλύτερη συνεργασία ανάμεσα στους εταίρους. Επίσης, ε, χρειάζονται ε, πιο αξιόπιστα δεδομένα, διότι χρειάζονται πιο έγκυρα στοιχεία για να μπορέσουμε να λαμβάνουμε σωστές ε, πολιτικές, ε, κοινωνικές ε, και περιβαλλοντικές αποφάσεις για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση οι εθνικές στατιστικές αρχές καταραίονται ότι έχουν πολύ περιορισμένους πόρους. Υπάρχουν όμως νέες ανάγκες για δεδομένα και συντονισμό σε εθνικό επίπεδο και αυτό πρέπει να συνδυαστεί με τα ξανόμενη πίεση για την εκπόνηση πιο έγκυρων εξόπιστων στοιχείων. Επίσης, συνειδητοποίησαμε όλοι πόσο δύσκολο είναι ε, να, ε, να έχουμε στη διάθεσή μας αρκετά ε, έγκυρα και αξιόπιστα αλλά και ταυτόχρονα διαφανή στοιχεία. Ε, το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα είναι το σύστημα, το μοναδικό σύστημα με μοναδικό στόχο να δίνει μια δομή για έγκυρα στοιχεία που θα μπορούν να χρησιμοποιούν όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτε, αλλά ταυτόχρονα και οι επιχειρήσει και οι ερευνητέ και οι ηθήνοντε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι απαιτούμενο ε, αυτό κομμάτι, απαραίτητο αυτό κομμάτι των εξελίξεων τη νέα ψηφιακή κοινωνία. Για να ενισχύσουμε περαιτέρω το σύστημα θα ήθελα, μπορώ, μπορώ να πω κι άλλα. Ένα λεπτό. Χρειάζεται τα εξή. των ε, ε, νέα στατιστικά εργαλεία και έχοντα κατά νου τη νέα οικονομική διακυβέρνηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, ούτω ώστε να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε του αρχικού στόχου. Κάτι που είναι αδύνατο εάν δεν είναι υψηλή ποιότητα και διαφανή τα στατιστικά στοιχεία. Ε, στα οποία βασίζονται οι αποφάσεις. Δεύτερον, χρειαζόμαστε ένα πολιτικό σύστημα ε, που θα υποστηρίζει με πόρους ε, το ευρωπαϊκό στατιστικό σύστημα. Ε, τον επόμενο μήνα ελπίζω να παραταθεί ε, το πλαίσιο λειτουργίας ε, του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος από το Κολέγιο των Επιτρόπων, από το Σώμα των Επιτρόπων, το οποίο κανονικά θα διαρκέσει μέχρι το 2020. Οπότε όλα τα συστήματα στα πλαίσια του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου μέχρι το 2020 θα καλυφθούν και από το νέο Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα. Χρειαζόμαστε πρικοδότηση για να υλοποιηθεί αυτή η εντολή. Υψηλή ποιότητα στατιστικών στοιχεία. Είναι μια επένδυση που θα κάνουμε και που ε, υποστηρίζει και η δική σας Επιτροπή, όπως αναφέρατε στη γνωμοδότησή σας για το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2016. Ε, περιμένουμε και την ε, μελλοντική σας πρόταση νομοθετικού χαρακτήρα για να υποστηρίξετε και να δώσετε συνέχεια σε αυτό το αρχικό σας ψήφισμα. Θα πρέπει λοιπόν να αντιληφθούμε ότι είναι ράχο κοκαλιά για τη λήψη σωστών αποφάσεων Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το νέο Ευρωπαϊκό Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα. Χρειάζονται μεταρρυθμίσεις, όμως ε, προτού γίνουν ε, βαθιές μεταρρυθμίσεις οποιοδήποτε σύστημα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, χρειάζονται ε, βαθιές μεταρρυθμίσεις στο Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα. Σας ευχαριστούμε κύριε Ράντερ Μάχερ, πολύ ωραία η παρουσίασή σα και φυσικά συμφωνούμε απολύτως ότι είναι μια επένδυση για το μέλλον τα κονδύλια που διοχετεύουμε στη μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος ο κύριος Μπουρχαμπάλης ο πρώτος ομιλητής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Ραντεμάχερ, χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Έχω δύο σύντομες ερωτήσεις. Η πρώτη αφορά αυτό το οποίο είπατε και πέρσι. Ίσως θυμάστε την τελευταία φορά που ήρθατε. Ετέθη το ζήτημα σε ποιο βαθμό οι εθνικές στατιστικές αρχές είναι ανεπηρέαστες από πολιτικές επιρροές. Μπορείτε να μας πείτε πώς αξιολογείτε την ε, κατάσταση σήμερα. Δεύτερον, κάτι που σχετίζεται με την κρίση χρέους. Αυτό το οποίο λέμε κάπως πιο διπλωματικά τις λεγόμενες στατιστικές ανακρίβειες που αφορούσαν ιδιαίτερα κάποιες χώρες που μας, απασχολούν, μας απασχόλησαν και φέτος. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Τα στατιστικά ιδιαίτερα όσον αφορά τις κρατικές δαπάνες και τα έσοδα έχουν ε, βελτιωθεί όσον αφορά την ακρίβειά τους και την αξιοπιστία τους έτσι ώστε να συνδυαστούν με άλλους παράγοντες όπως ε, η ανταγωνιστικότητα για να καταλήξουμε σε μια αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας των κρατών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, θα απαντήσω στα αγγλικά αν μου επιτρέπετε. Βεβαίω αντιλαμβάνω πως οι Γερμανοί συμπατριώτες θα ήθελα να μιλήσω γερμανικά. Να ξεκινήσω με δεύτερη ερώτηση η ποιότητα των στατιστικών στοιχείων. Βελτιώθηκε και βελτιώνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια. καθώς εξετάζουμε τις λεπτομέρειες σε συνδυασμό και σε συνεργασία με τις ελεγκτικές και στατιστικές αρχές. Η απόδειξη είναι πως ε, όποτε βρίσκουμε κάποια προβλήματα όπως στην περίπτωση της Βαλένθιας που ανέφερα ε, δόθηκε αμέσως συνέχεια και υπήρχε και ένα σήμα προληπτικό θα έλεγα. Οπότε υποθέτω πως παγκοσμίω ε, τα στατιστικά στοιχεία της γενικής κυβέρνησης είναι τα δυσκολότερα. Ελέγχονται πάρα πολύ εντατικά Υπάρχει ο μηχανισμός της Eurostat και λοιπόν και ένα περαιτέρω βήμα θα ήταν να εισαχθεί να εισαχθούν τα λεγόμενα έψας ε, τα ευρωπαϊκά λογιστικά πρότυπα του δημοσίου τομέα έτσι ώστε σε κάθε δήμο, σε κάθε νησί σε κάθε νοσοκομείο θα ήταν αναγκασμένα τα κράτη-μέλη να συμφωνήσουν στα ίδια λογιστικά πρότυπα για το δημόσιο. Ένα βαθμό συγκρισιμότητας που δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Κοιτάμε παραδείγματος χάρη μεγάλες συμβάσεις και τα λοιπά. Αλλά δεν μπορούμε να πάμε σε κάθε νησί. Αυτό λοιπόν ε, μας είπατε να εξετάσουμε το 2011. Είδαμε τις εκθέσεις. κάνουμε, σημειώνουμε καλή πρόοδο και μέχρι το 2020 είμαστε σε μια εθελοντική φάση και έτσι θα εισαχθούν σιγά σιγά κοινά λογιστικά πρότυπα για το δημόσιο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, η πολιτική επιρροή επί των εθνικών στατιστικών αρχών. Είδατε την επιθεώρηση από τους ομολόγους που γίνεται όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε χώρες όπως η Ισλανδία. Και πραγματικά βλέπουμε πολύ διάφανη αξιολόγηση της κατάστασης. Και αυτό είναι μοναδικό. Στο παγκόσμιο στατιστικό σύστημα δεν υπάρχει ένα συγκρίσιμος μηχανισμός ελέγχου που προλαμβάνει την πολιτική επιρροή. Τόσο πολύ. Σας ευχαριστώ κυρία Ελίζα Φερέιρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ που ήρθατε και χαρά μας που σας βλέπουμε. Αναφερθήκατε στην Ελλάδα. Είχαμε ρωτήσει λοιπόν τον κύριο Αλμούνια τότε υπεύθυνο και μας είπε ότι το 2004-2005 είχε αναφερθεί στην ποιότητα των ελληνικών στατιστικών στοιχείων και στην δυνατότητα ελέγχου από την Eurostat η οποία περιεκόπη για πολιτικούς λόγους. Τώρα θεωρείτε ότι έχετε την δυνατότητα αυτή για να ελέγξετε εις βάθος και να αξιολογήσετε την ποιότητα στατιστικών στοιχείων. Δεύτερον, όταν ε, εμείς ε, Ε, ως Επιτροπή επισκεφθήκαμε το 2008-2009 την Goldman Sachs μας είπαν πως αυτό που είναι με την Ελλάδα έγινε και με άλλα κράτη-μέλη και πολύ ισχυρά. Μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε πως υπάρχει η δυνατότητα και η ανεξαρτησία να δείτε όχι μόνο τις περιπτώσεις της Ελλάδας και της Ισπανίας αλλά και των πιο ισχυρών χωρών με τα ίδια μέτρα και σταθμά. Κατόπιν, ήμουν ε, εισηγήτρια στο θέμα των μακροοικονομικών ανισορροπιών και ο στόχος ήταν να αντιληφθούμε πώς λειτουργεί η Ευρωζώνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς αντιδρούν οι οικονομικές μεταβλητές στην κοινή αγορά και στους ε, κοινούς κανόνες. Γι' αυτό ακριβώς ε, Ήμασταν πάρα πολύ προσεκτικοί όσον αφορά τον πίνακα βαθμολογία, αλλά εντωμεταξύ η ανάλυση που γίνεται είναι αναχώρα. Δηλαδή ε, δεν είχε εντωμεταξύ νόημα ο πίνακα βαθμολογία. Μπορείτε λοιπόν να μας διαβεβαιώσετε πως ε, αυτή η διάχυση συστημάτων διαπεπλεγμένων θα διατηρηθεί όταν αξιολογείται και πάλι τους δείκτες του πίνακα βαθμολογίας. Τέλος, αυτό το οποίο αναφέρατε, ενημερώνεται τα κράτη-μέλη για την ανάγκη κάποιων διασφαλίσεων όταν συστήνεται περικοπέ προπολογισμού και διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει ότι κάποια σημεία τη δημόσια διοίκηση θα πρέπει να προστατευτούν, μεταξύ των οποίων και η στατιστική υπηρεσία. Γιατί αν μειωθεί η ποιότητα τη ε, στατιστική υπηρεσία, ε, τότε είναι δύσκολο μετά να έχουμε σωστέ ε, πληροφορίε. Ευχαριστώ. Okay, thank you very much. Ναι, ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Να απαντήσω με τη σειρά αν έχουμε αρκετές αρμοδιότητες ώστε να εμποδίσουμε το, όσα συνέβησαν ε, το 2004 να ξανασυμβούν. Τεχνικός, νομικός ναι, πολιτικός όχι. Στην Ελλάδα είναι σαφές ότι χρησιμοποιήσαμε όλες τις αρμοδιότητές μας ε, το 2010 τον Αύγουστο όταν η νομοθεσία που δεν είχε μεταγραφεί το 2005 έκλεισε. Έχουμε τώρα τη δυνατότητα να πάμε στα κρατη και να πούμε ναι, ανοίξτε αυτές τις πόρτες παρακαλώ, θέλουμε να ελέγξουμε τα βιβλία σας. Αυτό δεν ισχύσε. Όμως αυτό λειτουργεί μόνο αν έχουμε εταίρους επιτόπου, συνομιλητές που είναι αξιόπιστοι εταίροι. Αυτό συνέβη στην Ελλάδα, ίσχυσε στην Ελλάδα με τον πρόεδρο που ε, έληξε η θητεία του τον Ιούλιο. Και τώρα ξέρετε ότι είναι ενώπιον του δικαστηρίου επειδή ε, υπολόγισε τα στοιχεία με λάθος τρόπο. Χρειαζόμαστε ένα συνομιλητή και μια νοοτροπία στα κρατη που δεν είναι ε, εχθρική στις ε, ουδέτερες στατιστικές. Αν πιστεύεις ότι με έναν ε, τέτοιο υπολογισμό μπορείς να κάνεις αξιόπιστες στατιστικές, ε, τότε έχουμε πρόβλημα. Και αυτό το είναι πολιτικό πρόβλημα, δεν μπορούμε να το λύσουμε εμείς από την Eurostat. Εμείς πρέπει να έχουμε μια ατμόσφαιρα που να μας επιτρέπει να δουλέψουμε. Δεύτερον, στην Goldman Sachs ήμουν στην ακρόαση αυτή εδώ που αφορούσε τα swaps. Τα swaps στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Νομίζω πως για τα swaps λύσαμε το πρόβλημα μαζί με τα κράτη-μέλη, διότι έχουμε μία συμπεφωνημένη μέθοδο για το πώς καταγράφονται τα swaps. Έχουμε δηλαδή ένα εργαλείο επί του οποίου συμφωνούμε όλοι και συμφωνούμε όλοι πως έτσι θα πρέπει να λειτουργήσουμε. Αλλά βέβαια πάντοτε προσπαθούμε να προλάβουμε και τις νέες ιδέες του χρηματοπιστωτικού τομέα. Για το MIP θα πρέπει να πούμε ποιοι είναι οι βασικοί οι δείκτες και ποιοι είναι, ποιες είναι οι υπόλοιπες στατιστικές που τους στηρίζουν. Το θέμα του MIP είναι ένα θέμα με το οποίο ασχολήθηκε ήδη το προηγούμενο κοινοβούλιο και αυτό εξετάζει τους βασικούς δείκτες, την κορφή του παγόβουνου, τα λέγαμε. Με την έννοια ότι αν ελέγξουμε την ποιότητα αυτού του top επίπεδου έχει ένα είδος έμεσου ελέγχου. Αυτή είναι η λογική. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε το ίδιο επίπεδο ποιότητας για 250 στατιστικά προϊόντα, που είναι πάνω κάτω ο κατάλογος προϊόντων που έχουμε. Έχουμε δηλαδή προϊόντα όπως οι στατιστικές για τις υδατοκαλλιέργειες στρίδια, μύδια και σχετικές μετρήσεις. Και πρέπει να ε, κατανείμουμε το επίπεδο ποιότητα για αυτή τη συγκεκριμένη στατιστική. Αν πούμε ότι εκεί θέλουμε να έχουμε το ψηλότερο πεδίο, επίπεδο μάλλον ποιότητα, τότε θα πρέπει αυτό να το δεχτούμε. Αλλά δεν είναι πάντα το ίδιο. Για το MIP θα πρέπει να έχουμε full έλεγχο, πλήρη έλεγχο. Τώρα, πόροι στα κράτη-μέλη. Και αυτή θα είναι η τελευταία μου παρατήρηση. Και οι εθνικές επενδύσεις θα πρέπει να θεωρηθούν επένδυση. Επένδυση η οποία θα πρέπει να είναι ε, εκτός του πακέτου επενδύσεων. Μάλιστα chciałbym zadać pytanie dotyczące bilansu płatniczego. κύριε Διευθυντά, έχω μια ερώτηση για το θέμα του ισοζυγίου πληρωμών που είναι αυτή τη στιγμή στον τριμερή διάλογο και δεν έχουν επιληθεί κάποια ζητήματα. Πρώτα απ' όλα το θέμα των στατιστικών στοιχείων για τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Στο πλαίσιο του πραγματικού τελικού δικαιούχου πώς το ερμηνεύουμε αυτό, γιατί αντιλαμβάνομαι πως κάποια κράτη-μέλη αυτή τη στιγμή δεν συλλέγουν τέτοια δεδομένα και μάλλον πρέπει να το δούμε αυτό από την πλευρά των άμεσων ξένων επενδύσεων και των ε, μητρών επιχειρήσεων. Πότε θα πρέπει να περιμένουμε τα κρατη να αρχίσουν να συλλέγουν τέτοια δεδομένα. Ποιο είναι το βασικό εμπόδιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη συλλογή τέτοιων δεδομένων για τις άμεσες ξένες επενδύσεις ή άλλες ξένες επενδύσεις και πάλι δίνοντας βάρος στον πραγματικό τελικό ιδιοκτήτη. Και η δεύτερη μου ερώτηση, η διαφορά μεταξύ συναλλαγών που είναι πραγματικές νέες επενδύσεις σε αντίθεση με κάποιες εξαγορές. Πώς μπορούμε να κάνουμε αυτή την διάκριση. θεωρείτε πως ε, η πλήρης δημοσιοποίηση τέτοιων δεδομένων μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα σε μικρότερα κράτη-μέλη. Όταν ετησίως οι τέτοιες, τέτοιου είδους άμεσες ξένες επενδύσεις είναι πολύ μικρότερες, ενώ σε κάποια κράτη-μέλη δεν υπάρχει ακριβώς πλήρης δημοσιότητα για τον λόγο αυτόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις σας. Για την πρώτη ερώτηση η απάντηση είναι πως ε, τώρα κοιτάμε με τα κράτη-μέλη με ποιο βαθμό μέσω κάποιων πιλωτικών μελετών μπορούμε να λύσουμε το ζήτημα που αναφέρατε. Και η γενική άποψη είναι πως η πιλωτική αυτή μελέτη θα πρέπει να γίνει έτσι ώστε μέχρι το 2018 να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάποια μεθοδολογικά ορθή απάντηση. Και εδώ πέρα θα ήθελα να κάνω διάκριση μεταξύ των δύο τύπων συναλλαγών που αναφέρατε για τις πραγματικά νέες επενδύσεις. Αυτό διεθνώς δεν αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας. Οπότε θα πρέπει να το δούμε με τις πιλωτικές μελέτες και με τους εταίρους μας. Ε, το ισοζύγιο πληρωμών, όπως ξέρετε, βασίζεται σε κάποιες προδιαγραφές του ΔΝΤΑΦ. Οπότε πρέπει και εμείς και εσείς να βασιστούμε στην διεθνή συνεργασία, κατά το οποίο σημαίνει να συμφωνήσουμε με όλα τα κρατημέλη και με αυτά που έχουν ε, κάποια δυσκολία στο να μετρήσουν κάποια πράγματα. Και να συμφωνήσουμε βέβαια με τους εταίρους μας ε, στην Ουάσιγκτον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και σας κύριε Ραντεμάχερ. Δύο πράγματα έχω που θα ήθελα να συζητήσω μαζί σας. Το πρώτο το αναφέρατε. το ότι η Κομισιόν επέβαλε πρόστιμο στην Ισπανία και για το θέμα των στατιστικών στοιχείων της Βαλένθιας. Αυτό βεβαίω είναι λόγω των νέων αρμοδιοτήτων που έχει Κομισιόν με το ...και Ήταν η πρώτη τέτοια περίπτωση κυρώσεων για στατιστική απάτη και το ερώτημα είναι τι άλλα εργαλεία αναπτύσσεται αυτή τη στιγμή έτσι ώστε να υπάρξει σαφής ε, διάκριση μεταξύ σφάλματος και απάτης. Πρώτον. Δεύτερον, ποιο είναι το όριο, πώς κάνετε εσείς την αξιολόγηση. Και τρίτον, ποιες άλλες χώρες ή περιφέρειες εξετάζετε. Γιατί μιλάμε πάντα για τα κράτη-μέλη, αλλά βεβαίως όσο πιο βαθιά φτάνει κανείς, ε, τόσο περισσότερο συναντά συζητήσεις για ΣΔΙΤ, για το πώς οι Δήμοι ε, κάνουν τα λογιστικά τους τώρα ή τα έκαναν στο παρελθόν και βεβαίως ε, κοιτάγαμε μόνο στο εθνικό επίπεδο αλλά αν κοιτάξουμε πιο κάτω θα βρούμε και άλλα πράγματα. Δεύτερον, κάτι το δεν σχετίζεται με το πρώτο ζήτημα, είναι μια συζήτηση που υπάρχει σε πολλά κράτη-μέλη. Ο οικονομικός αντίκτυπος των δαπανών για την υγεία. Υπάρχουν σοβαρές αποκλήσεις στην διαχείριση των συστημάτων υγείας και είναι δύσκολο να συλλεχθούν αυτά τα στατιστικά στοιχεία, αλλά έχω την αίσθηση πως ε, ειδικά σήμερα θα μπορούσαμε έτσι να διαμορφώσουμε τις πολιτικές στα, στα κράτη-μέλη για να δούμε πώς ακριβώς θα τα χρήματα για την υγεία. Σας ευχαριστώ για την πρώτη σας ερώτηση. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε διαχωρίσει την απάτη από την εσκεμμένη λάθος ε, πληροφόρηση. Κάτι το οποίο θα πρέπει να γίνει βεβαίως όταν θα πρέπει να κάνουμε την διάκριση. Όμως η διαδικασία της ε, Βαλένθιας ε, περιέλαμβανε και βοήθεια από τον Όλαφ, ε, την υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης. Οπότε, κοιτάξτε, επειδή εμείς οι στατιστικολόγοι δεν έχουμε και τα εργαλεία στην διάθεσή μας για να κάνουμε έρευνα. Οπότε το διαχειριστήκαμε σαν να ήταν υπόθεση απάτης και η διαδικασία νομίζω ήταν ε, οπωσδήποτε περίπλοκη. Τώρα βασιζόμαστε πάρα πολύ στις ελεγκτικές αρχές, τις ανώτατες ελεγκτικές αρχές των κρατών μελών. Και στη Βαλένθια και σε άλλες ε, περιπτώσεις ε, παίρνουμε τις πληροφορίες από τις αναφορές ελέγχου. Και στην Βαλένθια το ίδιο συνέβη. Η τοπική ελεγκτική αρχή το είχε επισημάνει. Και αυτή ήταν η αφετηρία. Είχαμε στενή συνεργασία και με το, δικαστή, το ελεγκτικό συνέδριο. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο συνεργάζεται με τα Εθνικά Ελεγκτικά Συνέδρια και αυτός είναι ο τρόπος μας ε, με τον οποίο προσπαθούμε να λύσουμε το πρόβλημα. Συνεργαζόμαστε λοιπόν με τις ελεγκτικές αρχές ε, στα κράτη-μέλη. Τώρα για το θέμα της υγείας και την ποιότητα των δεδομένων. Μπορούμε να πούμε πως σε πολλές ε, τέτοιες ε, περιπτώσεις η αφετηρία ήταν ο τομέας της υγείας. Στην Ελλάδα και στην Βαλένθια παραδείγματος χάρη όπου ήταν λανθασμένες οι αναφορές. Ο κλάδος λοιπόν αυτός είναι προφανώς ο πιο ευπαθής θα έλεγα για τέτοιου προβλήματα. Το γνωρίζουμε αυτό. Γι' αυτό ακριβώς δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή όποτε πάμε στα κράτη-μέλη με τους επιθεωρητές θα έλεγα. για να δώσουμε βάρος ε, στον τομέα της υγείας. Ευχαριστώ. Η απόφαση του Συμβουλίου για τα 18 εκατομμύρια νομίζω ε, χαρακτηρίζεται ως ε, εξαιρετικά πλήμελης. Σβέν Γίγκολντ. Ευχαριστώ. Κύριε Καλώς ήρθατε και πάλι στην μικρή και εκλεκτή επιτροπή μας. Να θέσω δύο ερωτήματα. Το ένα το έχω ξαναβάλει και άλλη φορά. Στο σημείο 4.3 το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Πρόγραμμα αναφέρεται σε στην απέτηση του Κοινοβουλίου για να κάνει περισσότερα η Eurostat για να φανεί η οικονομική συνεισφορά των κοινωνικών φορέων. Τι έχετε κάνει στο μέτωπο αυτό. Δεύτερον, ένα αγαπημένο δικό μου θέμα το ότι δεν καλύπτονται στρατηγικά εις δίτ, οι συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και η τάση των κρατών μελών λόγω του περιορισμού του ΣΥΞΠΑΚ να κάνουν διάφορους κρυφούς προϋπολογισμούς. Τώρα διαβάζω 10 Φεβρουαρίου φέτος για πρώτη φορά μιλήσατε για αυτούς τους σκιώδεις προϋπολογισμούς ε, μεταξύ των οποίων και της ε, ΣΔΙΤ και εκεί πέρα λέτε πως στη Γερμανία δεν υπάρχουν ε, μας λένε πως δεν υπάρχουν στη Γερμανία καθόλου εκκρεμότητες από ΣΔΙΤ λίγο απίθανο αυτό γιατί δεν ξέρουν καν οι δήμοι ποιε είναι οι εκκρεμότητες. Όλοι ξέρουν πως και αυτοί που λαμβάνουν τις αποφάσεις δεν έχουν ιδέα για το τι κινδύνους αναλαμβάνουν. Αναρωτιέμαι λοιπόν πόσο έχετε προχωρήσει όσον αφορά τις κυρώσεις ε, απέναντι στη Γερμανία ειδικά που αντιστάθηκε στο να καλύπτονται αυτά τα πράγματα στα στατιστικά στοιχεία και να σας πω ε, αν δεν εμπιστευόμαστε την Γερμανία θα ήθελα να μάθω πόσο αξιόπιστα βρίσκεται αυτά τα στοιχεία γενικότερα και τι σκοπεύετε να κάνετε για να υπάρχει πλήρης διαφάνεια στους κοιόδους προπολογισμούς. Δεν είναι δυνατόν να κλείνουμε μια τρύπα και κάποιοι άλλοι να ανοίγουν κρατήρες. Ευχαριστώ. Αρχίσαμε το πρώτο σας ερώτημα. Ναι, Όντως, ε, μας ζητείτε να ερευνήσουμε τέτοιους τομείς, όπως η ΣΔΙΤ, παραδείγματος χάρη. Όμως, για να είμαι ειλικρινέστατος μαζί σας, περιορίστηκαν πάρα πολύ τα αποτελέσματα που είχαμε, διότι δεν είχαμε αρκετούς πόρους. Δεν μπορέσαμε στην ουσία να έχουμε πρόοδο. Συζητήσαμε με τα κράτη-μέλη διάφορες προσεγγίσεις, μεν, όμως ε, είναι τόσο τραγική κατάσταση στα κράτη-μέλη σε σχέση με τους πόρους που έχουν οι εθνικές στατιστικές αρχές ε, ώστε δεν μπορούμε να είμαστε ούτε καν σίγουροι ότι εκπληρούνται οι νόμιμες, ε, οι βάσει του νόμου υποχρεώσεις που έχουν τα κράτη-μέλη. Ακόμη και για τα προβλεπόμενα δεν φτάνουν οι πόροι. Ο κύριος Κίκολ, ναι, κατάλαβα ότι δεν, είσαστε σε θέση, δεν είναι σε θέση τα κράτη-μέλη να εκπληρώσουν αυτές τις υποχρεώσεις ε, λόγω περιορισμένων πόρων, όμως επανέρχομαι και σε σχέση με αυτά που είπατε στην αρχική σας παρουσίαση, ε, τα ευρωπαϊκά στατιστικά προγράμματα είναι επίσης ε, υποχρεωτικά. Δεν καταλαβαίνω ποια είναι υποχρεωτικά και ποια όχι βάσει αυτών που μας λέτε. Είναι τραγικά αυτά που μας λέτε ουσιαστικά. Τι εννοείτε. Απάντηση. Έχουμε κάποιους πόρους για να σημειώσουμε πρόοδο σε αυτό το τομέα, όμως χρειαζόμαστε στατιστικά στρώματα τα οποία δεν ρυθμίζονται λεπτομερώς νομοθετικά. όπως μελέτες που θα χρειαζόμασταν για να έχουμε τις βασικές πληροφορίες. Δηλαδή δεν είναι τμήμα του στατιστικού και εκτιμένου και γίνεται σε θελούσια βάση από τα κράτη-μέλη μόνο. Άλλες συνιστώσεις δεν συντρέχουν και γι' αυτό προσπαθούμε να συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη για να βρούμε μια λύση. Αυτό είναι μέλο, μέρος συγγνώμη, του πακέτου προτάσεων που θα καταθέσουμε το 2016 για τις μελέτες ε, βάσει του επωνομαζόμενου Ευρωπαϊκού Ενωπαϊμένου Κανονισμού για τις μελέτες για τα κοινωνικά ε, ζητήματα και εκεί θα δείτε κάποιους παραμέτρους που δίνουν εν μέρει απάντηση, απάντηση σε αυτό το ζήτημα. Έχουμε δηλαδή δραστηριοποιηθεί και σε αυτό το τομέα. Όμως δεν έχουμε φτάσει στο σημείο όπου θα μπορούσαμε να σας δώσουμε ε, αυτά αποτελέσματα. Είμαστε σε φάση ανάπτυξης. Αυτές οι μελέτες ε, για τα νοικοκυριά ε, θα τις κάνουμε στα πλαίσια του κανονισμού για τις κοινωνικές στατιστικές. Και εποδηποτάσουμε στο 2016. Τώρα, για την καταγραφή των ΣΔΙΤ, Οι γερμανικές αρχές μας είπαν πως όλες οι ΣΔΙΤ καλύπτονται. Τι σημαίνει αυτό. Οι ΣΔΙΤ που είναι γνωστές σε επίπεδο ομοσπονδιακό και κρατηδίων. Ε, σε δημοτικό επίπεδο Όμως πρέπει να δοθεί μια απάντηση και σας είπα ότι τα ευρωπαϊκά λογιστικά πρότυπα κανονικά πρέπει να έχουν εισαχθεί. Αυτά πρέπει να υιοθετηθούν κύριος Γίγκολ. Δηλαδή είναι πλημελή τα στοιχεία γιατί οι περισσότερες ΔΙΤ είναι σε δημοτικό επίπεδο. Ε, τότε πείτε μου πότε θα χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία που έχετε στη διάθεσή σας τόσο ώστε να παίρνετε σωστές στατιστικές από τη Γερμανία για αυτά τα ζητήματα. Εάν τελικά δεν καλύπτονται είναι ε, τα, τα μηδενικά στατιστικά στοιχεία πλημελή. Αυτό εννοείται. Καλά κατάλαβα. Απάντηση. Όχι έχουμε πάρει μια κοινοποίηση από τις γερμανικές αρχές που λένε ότι οι ΣΔΙΤ καλύπτονται 100%. Στις, ε, στην κοινοποίηση που μας κοινοποιεί η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση για τα οικονομικά της στοιχεία. Υπάρχουν ε, λοιπόν κάποιες ΣΔΙΤ που δεν καλύπτονται, ε, εκτός και αν δεν υπάρχουν ΣΔΙΤ σε δημοτικό επίπεδο. Καλά καταλαβαίνουμε. Είναι μια τρύπα αυτή. Θα δοθεί συνέχεια σε αυτό. Ευχαριστώ και θα μιλήσω Ολλανδικά και για τις ΕΣΔΙΤ. Κοιτάξτε, στο Βέλγιο ανησυχεί ιδιαίτερα το τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Είναι βεβαίως ένα ζήτημα το οποίο συζητάμε εδώ και χρόνια και το ερώτημα είναι αν θεωρείτε ότι τα κριτήρια τα οποία χρησιμοποιούν, χρησιμοποιεί η μπορεί να καλύψουν τις ΣΔΙΤ και ειδικά βεβαίως την απόκληση από τον κόσμο των επιχειρήσεων όπου οι επενδύσεις ε, σε πάγια καλύπτονται διαφορετικά. Και μια προσωπική ερώτηση υφίσταται το πρόβλημα αυτό και σε άλλες χώρες ή αφορά μόνο τις ε, βέλγικες ε, ΣΔΙΤ οι οποίες από ό,τι φαίνεται δεν συμβάζονται πάρα πολύ με το ευρωπαϊκό πρότυπο. Ε, για να αρχίσω από Την διευκρίνηση. Οι κανόνες που εφαρμόζουμε για την καταγραφή των ΣΔΙΤ σε όλα τα κράτη-μέλη είναι οι κανόνες που ισχύουν και νομοθετήσατε εσείς. Λέγεται ΕΖΑ, το Ευρωπαϊκό Λογιστικό Σύστημα. Ε, το ΕΖΑ 2010 είναι αυτό το οποίο ακολουθούμε σε αυτή την περίπτωση. Και το εφαρμόζουμε αδιακρίτως ανεξαρτήτως του ποιο είναι το κράτος μέλος. Και βέβαια για το Βέλγιο η πυκνότητα των ΣΔΙΤ και η δυσκολία είναι θα έλεγα αν μου επιτρέπετε δυσανάλογη. Αλλά οι κανόνες ε, είναι οι συνήθεις ε, κανόνες ε, όσον αφορά την λογιστική με βάση τα δεδουλευμένα. Δηλαδή, αν η γίνεται με έναν τρόπο ώστε τον κίνδυνο τον λαμβάνει το δημόσιο και ληφθεί μια απόφαση από το δημόσιο, τότε είναι δημόσιο. Αυτά λένε οι αρχές ε, του λογιστικού. Και έχουμε επενδύσει πολύ χρόνο στην καλύτερη επικοινωνία τα είχαμε συζητήσει και με τους Βέλγους εταίρους μας συγκεκριμένα πρέπει να έχουμε κατά νου πως εμείς είμαστε το δεύτερο επίπεδο θα έλεγα συζήτησης δεν είμαστε ρυθμιστικές αρχές. Οι εθνικές αρχές, δηλαδή η Στατιστική Υπηρεσία και η Βελγική Κεντρική Τράπεζα, είναι αυτές που κάνουν τον διάλογο αυτόν. Βεβαίως εμείς ευχαρίστως να βοηθήσουμε, αλλά είμαστε στο παρασκήνιο θα έλεγα, σε μια δεύτερη φάση. Βεβαίως έχουμε και την επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και ελπίζω τελικά η επένδυση αυτή να αποδώσει με καλύτερη κατανόηση των κανόνων μας και των νομικών αρχών. Ευχαριστώ Νίνα Τζιλ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε και για την ε, παρουσίασή σας. Ε, νομίζω πως ε, αποφάσεις που βασίζονται σε στοιχεία πραγματικά θα μας βοηθήσουν εμάς τους νομοθέτες για να δούμε αυτές τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Το πρόβλημα είναι ακριβώς να έχουμε έγκαιρες πληροφορίες. Αν δούμε π.χ. το ζήτημα το προσφυγικό. Το βασικό πρόβλημα είναι το να έχουμε ακριβείς πληροφορίες. Αν δούμε δε και τις ε, δικές σας εκτιμήσεις, ε, μιλάμε για 750.000 άτομα μέχρι στιγμής φέτος, αλλά είναι ασαφές ε, γιατί τα κριτήρια που χρησιμοποιείται είναι οι άνθρωποι που ζητάνε άσυλο που είναι γύρω στους 700.000. Υπάρχουν όμως πολλοί που ήρθαν και δεν ζητάνε άσυλο και με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έφτασαν και ήρθαν εδώ. Δεδομένη της πολιτικής σημασίας ε, του να είναι σωστά αυτά τα δεδομένα, πώς μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να βασιστούμε σε αυτά τα στοιχεία, γιατί το τίμημα μπορεί να είναι πάρα πολύ υψηλό αν δεν έχουμε σωστές πληροφορίες. Είτε το να ψηφίζει ο κόσμος ε, ακραία κόμματα ή ε, και από το Ηνωμένο Βασίλειο θα επηρεάσει το δημοψήφισμα ας πούμε. Μπορείτε λοιπόν να μας πείτε μέσω μακροπρόθεσμα το ποιες είναι οι οικονομικές συνέπειες του φαινομένου σε σχέση με την εθνική αγορά εργασίας, τους προϋπολογισμούς και τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. Ένα άλλο ξεχωριστό ζήτημα. Ε, λέμε πως τα ευρωπαϊκά στατιστικά στοιχεία δημοσιεύονται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι περιφερειακές διαφορές. Υπάρχουν μεγάλες κοινωνικο-οικονομικές διαφορές μεταξύ Λονδίνου και της υπόλοιπης χώρας. Πώς μπορούμε να τις δούμε αυτές. Στα στοιχεία της Γιώργης, ευχαριστώ. Mm. Σας ευχαριστώ. Να αρχίσω με την πρώτη πολύ πολύ δύσκολη ερώτηση, <clears throat> γιατί όπως γνωρίζουμε, το θέμα το προσφυγικό ήταν υπό εξέλιξη τους τελευταίους μήνες και μάλιστα με πολύ δυναμικό τρόπο εξελισσόταν. Και αυτό δεν μπορούσαμε να το έχουμε προβλέψει. Στην το μηχανισμό μας με έναν σωστό τρόπο. Αυτό που μπορούμε να προσφέρουμε για τους πρόσφυγες λοιπόν είναι ε, να έχουμε πληροφορίες για την μετανάστευση, την κινητικότητα της αγοράς εργασίας και ε, τα στοιχεία που συλλέγει η Frontex και άλλες αρχές, καθώς και οι αρχές ε, ασύλου. Αλλά ποτέ δεν θα είμαστε απόλυτα ενήμεροι μέχρι την τελευταία στιγμή, δηλαδή, για τις αφήξεις και τους ετούντες άσυλο, αν δεν έχουμε τις κατάλληλες πληροφορίες. Ε, το γεγονός ότι μπορούμε τώρα να έχουμε ε, τριμηνιαία στοιχεία με ένα μάξιμο ε, χρονικό κενό τριών μηνών, καθυστέρηση τριών μηνών, είναι ήδη πολύ καλή προσέγγιση της πραγματικότητας. Τώρα όσον αφορά τις οικονομικές επιπτώσεις για την αγορά εργασίας κτλ. Εκεί έχουμε συνεργασία στενή με την ε, ε, Γενική Διεύθυνση για την Απασχόληση, για την ε, Εσωτερικών και Οικονομίας. Και γιατί αυτοί έχουν τα καλύτερα εργαλεία, μπορούν να διακρίνουν ανάμεσα στα στοιχεία, τα στατιστική, τις στατιστικές και τα μοντέλα που υπολογίζουν τις πολιτικές επιπτώσεις. Εδώ λοιπόν έχουμε συνεργασία με τις υπηρεσίες της Κομισιόν. για τις περιφερειακές διαφορές. Συνεργαζόμαστε στενά με τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Ρέτζιο. Δεν ξέρω αν είδατε το yearbook, το, την επετηρίδα. Η περιφερειακή κατανομή, ιδιαίτερα όσον αφορά την αγορά εργασίας, και τέτοιου είδους στοιχεία, είναι ήδη αρκετά προηγμένη. Ωστόσο, αυτό που προσπαθούμε τώρα να κάνουμε είναι να επιταχύνουμε το την κοινωνική πτυχή και να έχουμε και βαθύτερες κατανομές περιφερειακές ε, συνδυάζοντας τις στατιστικές με γεωγραφικά στοιχεία και έτσι βελτιώνοντας τα μοντέλα εκτίμησης. Και... Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, προσπαθώντας να συνδυάσουμε τα κοινωνικά στοιχεία με την μακροοικονομία. Σας ευχαριστώ. Brian Hayes. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ εσάς και τους συναδέλφους σας που είστε σήμερα εδώ. Εγώ καταλαβαίνω πολύ πόσο δύσκολη είναι η εργασία σας ε, δεδομένης της σημασίας των στατιστικών που εκπονείτε και της ανεξαρτησίας που είναι τόσο σημαντική. Ε, έχετε ζωτικό ρόλο λοιπόν να παίξετε και το αναγνωρίζω αυτό. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση για τη σύγκριση επιδόσεων. Ε, στη χώρα μου στην Ιρλανδία από ό,τι κατάλαβα μια τέτοια έκθεση έγινε ο Μάρτιο φέτος και μετά υποβλήθηκαν 16 συστάσεις. Ποια συνέχεια δίνεται αναχώρα σε αυτές τις ε, συστάσεις. Μια τέτοια, ένας τέτοιος έλεγχος τι κάνετε. Πάτε, βλέπετε τι είναι καλό, τι είναι κακό, το ονοματίζετε και μετά πάει και τελείωσε ή υπάρχει κάποια συνέχεια. Γιατί Υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε ένα, μια ευρωπαϊκή προδιαγραφή, υπάρχει χώρος για βελτίωση, πρέπει αυτό να γίνει μετά. Μετά έχετε ένα κατάλογο για τις διαφορές που υπάρχουν και ισχύουν στις ευρωπαϊκές στατιστικές πληροφορίες και τη μεθοδολογία που έχει χρησιμοποιηθεί για να ε, φτάσουμε σε αυτές τις, πληροφορίε τις πληροφορίες και τον υπολογισμό αν ας πούμε πάρουμε τον τομέα των προεκβολών πληθυσμών, εξακολουθεί να υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις μεθοδολογίες των κρατών μελών και τη μεθοδολογία που χρησιμοποιεί η Eurostat. Έχουμε έναν οριστικό κατάλογο. Αν δεν το έχετε μαζί σας, μπορώ να τον έχω. Γιατί είπα να θα με ενδιαφέρε να δω ποιες είναι οι διαφορές που παραμένουν. Το ίδιο επιχείρημα ισχύει και για το απόδοση. Οι οικονομίε μας είναι πιο επιστιασμένε στις εξαγωγέ. Μπορείτε να το υπολογίσετε με ακρίβεια ή δεν ξέρουμε ακριβώς πόσο είναι το ΑΕΠ. Υπάρχει ένας συγκεκριμένος ορισμός και τέλος έχουμε κοινά στάνταρ για την σκιώδη οικονομία. Γιατί ανάλογα με το ποια είναι η φορολογία ε, στην οικονομία μας, αυτό επηρεάζει και την απόδοση της χώρας μας. Εξακολουθεί να υπάρχει σκιώδης οικονομία, μαύρη οικονομία, πώς την υπολογίζουμε, πώς την προσθέτουμε στο εθνικό ΑΕΠ και πώς τη λαμβάνετε υπόψη εσείς στις στατιστικές. Ευχαριστώ. Um, thank you very much. Uh, let me start with... εγώ σας ευχαριστώ. Όσον αφορά τη σύγκριση επιδόσεων και τις 26 ε, συστάσεις για την Ολλανδία και κατά πόσο θα δοθεί συνέχεια. Ναι, δίνεται συνέχεια η οποία γίνεται από εμά τη Eurostat. Η διαδικασία είναι ότι του χρόνου θα εκδώσουμε μια συνοπτική έκθεση που πάει στο Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα το Φεβρουάριο και μετά αυτή στέλνεται σε εσά και στο Συμβούλιο. Θα δείτε δηλαδή μια γενική εικόνα, μια γενική απεικόνηση. Και μαζί με τα κράτη-μέλη, στόχος είναι αυτός, να υπάρχει συνέχεια, να δίνεται συνέχεια. Βέβαια υπάρχουν συστάσεις και συστάσεις. Υπάρχουν αυτές που είναι πιο κρίσιμες και λιγότερο σημαντικές. Αυτές οι συστάσεις που συνδέονται με νομικές υποχρεώσεις, για παράδειγμα, να εφαρμοστεί ο κανονισμός 223, βεβαίως αυτές παρακολουθούμε με πολύ μεγαλύτερη προσήλωση και αφοσίωση. Και πιο αυστηρά από ό,τι άλλες συστάσεις που στόχο έχουν τη βελτίωση της ποιότητας. Εγώ θα έκανα τη διάκριση ανάμεσα σε minimum standard για τις στατιστικές οι οποίες είναι νόμιμες και νομοθετημένες σε πάση περιπτώσει και τις καλύτερες πρακτικές που είναι και ως κατευθύνσεις γραμμές. Για παράδειγμα προς μίμηση. Αυτό λοιπόν το παρακολουθούμε εμείς. Τώρα, κοινέ προδιαγραφές. Ναι, ξέρω πως υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις στην Ιρλανδική και στην Ευρωπαϊκή εκβολή που έχει δημιουργήσει μια, μια δυσαρέσκεια. Πάντως δουλεύουμε πάνω σε αυτό και Θέλουμε αυτό να το κάνουμε ετησίως όσον αφορά τις προεκβολές πληθυσμού. Ετησίως λοιπόν με, όπως κάνουμε και για όλες τις άλλες στατιστικές, με κοινά συμπεφωνημένες προδιαγραφές και κατευθύνες γραμμές για να ξεπεραστεί αυτό το δίλημα. Αυτό σημαίνει όμως ότι δεν θα έχουμε απαραίτητο ομοφωνία. Θα μπορούσε δηλαδή να συμβεί και στο μέλλον η Ιρλανδία να επιλέξει να χρησιμοποιήσει μια άλλη προεκβολή πληθυσμού και αυτό να μην είναι το ίδιο που έχουν συμφωνήσει οι άλλες χώρες μέλη. Χώρες μέλη. Τώρα, σκιώδης οικονομία μαύρη οικονομία. Αυτό είναι μια ερώτηση που ακούω τακτικά, συχνά πυκνά. Και ίσως να μπορώ να επαναλάβω αυτό που είπα και την προηγούμενη φορά, ότι δηλαδή μπορούμε να το διερευνήσουμε. Αυτό συνδέεται στενά και με κάτι που λέγεται παράνομες δραστηριότητες. Αυτές είναι οι ακραίες περιπτώσεις ανάμεσα σε συναλλαγές που μπορούμε να μετρήσουμε και να διακρίνουμε και αυτές που δεν μπορούμε. Και πρέπει να τις εκτιμήσουμε. Για τις παράνομες δραστηριότητες έχουμε συμφωνήσει με τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιούμε μια στάνταρ μεθοδολογία πέρυσι και αυτό ήταν σημαντικό για το GNI, για το εγχώριο καθόριστο προϊόν. Θυμάστε πέρσι έγινε λίγο ξεσηκωμός όταν τα νέα στάνταρ οδήγησαν σε ψηλότερα ΕΠΑ, Καθάριστο εγχώριο προϊόν. εκεί σε αυτές τις νέες προδιαγραφές είχαμε και ένα κομμάτι που ήταν οι παράνομες αυτές τις δραστηριότητες, ακόμα και αν ήταν πολύ μικρό το ποσοστό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τζάνι. Ζάνι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Γενικέ, θα ήθελα να ε, ρωτήσω δύο συγκεκριμένες ε, παρατηρήσεις ε, σε σχέση με κάτι που ήδη αναφέρθηκε. Η μία μου ερώτηση αφορά τις στατιστικές περί απασχόλησης. Μάλιστα έχω πολύ μεγάλες δυσκολίες να εξηγήσω στους ψηφοφόρους μας και στους εκλογεί στην Ουγγαρία πώς οι διάφορες ώρες εργασίας, οι μήνες, οι εβδομάδες κτλ. υπολογίζονται και θεωρούνται πλήρης απασχόληση. Ξέρω πως υπάρχουν τεχνικές προδιαγραφές και το καθεξής, αλλά είναι τόσο χαλαρά όλα αυτά που ένα απλός άνθρωπος δεν μπορεί να το συλλάβει. Δεν θεωρεί ότι κάποιος απασχολείται πλήρως, ενώ όταν δεν απασχολείται πλήρως, για παράδειγμα, κάποιες συμβάσεις που έχουμε σε κάποιες χώρες. Ε, σκοπεύετε να διευκρινίσετε κάπως περισσότερο ή να προσαρμόσετε το σύστημα στη ζωή, στην πραγματική ζωή. Στη χώρα μου τώρα την Ουγγαρία επίσης η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία αρνήθηκε να, να συλλέξει στατιστικές για την φτώχεια. Αυτό σημαίνει πως οι Ούγγροι δεν μπορούν να έχουν πληροφορίες σχετικά με τα επίπεδα φτώχειας σε, μια, σε αυτή τη χώρα, ενώ η κυβέρνηση δίνει συμβάσεις για σε κόσμο για 150 ευρώ το μήνα, που είναι ντροπή και δεν τα καλύπτει αυτά καμία στατιστική. Δεν μπαίνουν σε καμία στατιστική μέσα σε όλο αυτό το μηχανισμό όλα αυτά. Σας ευχαριστώ. Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Όσον αφορά τις στατιστικές απασχόλησης. Είναι κάτι που και εγώ το άκουσα όταν, όταν δούλευα ακόμα για τη Γερμανική Στατιστική Υπηρεσία, ότι οι ορισμοί σπόρο απέχουν από τις κανονικές λογικές ε, ε, αντιλήψεις. Ε, όμως οι ορισμοί είναι διεθνή στάνταρ του Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασίας. Εφαρμόζουμε λοιπόν αυτές τις προδιαγραφές που είναι διεθνώς συμπεφωνημένες. Εμείς τώρα επενδύουμε πολύ στο να προσθέσουμε συνιστώσεις ή πληροφορίες που θα μας επιτρέψουν στη συνέχεια να κάνουμε μια εκτίμηση, μια προσέγγιση και να μπορέσουμε να καλύψουμε το κενό ανάμεσα στην διεθνώς επιφωνημένη προδιαγραφή και την καθημερινή την αντίληψη του απλού κόσμου. Όταν ας πούμε εισήχθη το ευρώ, θυμάμαι ότι η σύζυγός μου μου είπε ναι, αλλά αυτά που μετράτε είναι τελείω τρελά, γιατί εγώ ξέρω καλύτερα τι τρέχει, γιατί ε, ότι η αγοραστική μου δύναμη, άρα ο πληθωρισμός είναι πολύ ψηλότερος. Η αγοραστική μου δύναμη έχει μειωθεί. Προσπαθώ λοιπόν, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να εξηγήσουμε καλύτερα, να χρησιμοποιήσουμε επιπλέον πληροφορίες. Για παράδειγμα, πριν μια εβδομάδα για πρώτη φορά δημοσιεύσαμε τις εισρωές και εκροές διαφόρων κατηγοριών από την αγορά εργασίας. Δηλαδή, άνεργοι, εργαζόμενοι, οι ζητούντες εργασία και οι υπόλοιποι. Αυτό προσπαθούμε τώρα να το κάνουμε συγκυριακά, αλλά πραγματικά προσφέρω τις υπηρεσίες μας για να σας βοηθήσω πέρα από το προϊόν που έχουμε, δηλαδή έχουμε και υπηρεσίες για να σας βοηθήσουν. Δεύτερον, επίπεδα φτώχειας. Ναι, πολύ δύσκολο θέμα σχετική φτώχεια με βάση την κατανομή του εισοδήματος. Στο να φτάσουμε σε πιο περίπλοκες μορφές φτώχειας, εδώ πρέπει να πω ότι είναι, ότι είναι από τα κύρια στοιχεία για το προγράμματό μας για τα επόμενα χρόνια είναι να επενδύσουμε μαζί με τα κράτη-μέλη και την Ουγγαρία δηλαδή μαζί ώστε να έχουμε συγκρίσιμες μετρήσεις κατανάλωσης εισοδήματος και πλούτου. Θέλουμε δηλαδή να γνωρίζουμε τις ανισότητες, όλο το φάσμα των ανισοτήτων και βελτιώνονται διερκώς οι γνώσεις μας. Είναι μία από τις ψηλότερες μας προτεραιότητες για τα επόμενα χρόνια. Σας ευχαριστώ, Μάρκο Βάλι. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εγώ έχω μια ευθεία άμεση ερώτηση. Οι στατιστικές ενδείξει που φτάνουν όσον αφορά όλη την Ευρώπη αλλά και για κάθε χώρα μετά μπορούν να ε, στηρίξουν ε, συγκεκριμένα είδη πολιτικών, δηλαδή ε, δημοσιονομικών ή νομισματικών. Γιατί, Γιατί οι επιχειρήσεις από τη στιγμή που βλέπουν μια και ένας και κόσμος μάλλον από τη στιγμή που βλέπουν θετικό ή αρνητικό πτώσιμο θεωρούν ότι τάδε πολιτική λειτουργεί. Το θέμα είναι κατά πόσο μπορούμε να εμπιστευτούμε αυτά τα στατιστικά στοιχεία τη, φάση, τη στιγμή που τροποποιούνται όπως έγινε το 2010 με την ε, ένταξη της ε, παράνομης οικονομίας και της μαύρης οικονομίας. Με αυτή την αναθεώρηση που έξι χρόνια μετά τη Λισαβόνα έγινε όσον αφορά τους στατιστικούς δείκτες για τον ε, πληθωρισμό. Δεν υπάρχει ο κίνδυνος ενός στατιστικού ντοπαρίσματος. Από την άποψη ότι δηλαδή έτσι στηρίζονται και δικαιολογούνται, αιτιολογούνται νομισματικές και δημοσιονομικές πολιτικές που διαφορετικά δεν θα έστεκαν. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Um, Πολύ σας ευχαριστούμε. Στατιστικό ντόπινγκ. Εμείς είμαστε λοιπόν η αρχή που καταπολεμεί το ντόπινγκ. Αυτό είναι ο ρόλος μας. Με το που αρχίζετε να χρησιμοποιείτε στατιστικά στοιχεία για να πάρετε αποφάσεις, τότε, όπως ο Τσαρλ Γκούτχαρτ έλεγε στον Ηνωμένο Βασίλειο, ο οικονομολόγος, με το που χρησιμοποιείτε δίκτυ για, την, ε, για να πάρετε αποφάσεις, αποδεικνύεται ότι είναι καλός δείκτης αυτός που χρησιμοποιείτε. Για να ε, σταματήσει αυτός ο φαύλος κύκλος, ε, αποφασίσαμε να έχουμε αυτή την νέα Δηλαδή, να είναι πιο ε, δυνατής οι στατιστικές αρχές, ε, πιο υγιείς. Προσπαθώ να σας πείσω ότι το ε, πιο εύρωστο ε, σύστημα που μπορεί κάποιος να έχει είναι το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα οι συνομοθέτες μας βοήθησαν να συγκροτήσουμε αυτό το νέο σύστημα. Ε, η αρχή και το τέλος, οτιδήποτε ε, προσπαθούμε να κάνουμε με τις ευρωπαϊκές στατιστικές βασίζεται στην εμπιστοσύνη. Ευχαριστούμε η Ιβάνα Μαλέτ. Ευχαριστούμε. Καλώς ήρθατε. Μιλήσατε για διαφάνεια και την αξιοπιστία των στατιστικών ε, δεδομένων. Είπατε ότι χρειάζονται και έλεγχοι σε εθνικό επίπεδο για την αξιοπιστία των στατιστικών αρχών. Τι όμως, ποιος αποφασίζει ε, γιατί πρέπει να γίνει ε, ο έλεγχος ε, και πώς θα υποβληθούν τα στοιχεία πάλι σε εθνικό επίπεδο γίνονται αυτό ή εσείς λαμβάνετε τα στοιχεία για να ολοκληρώσετε τον έλεγχο ή μόνο αν διαπιστωθεί παρατυπία θα πάει στο, κατευθείαν στο γραφείο του εισαγγελέα για να το διερευνήσουμε. Κατόπιν, ε, μιλήσατε για την ΕΚ και ξέρω ότι λειτουργείτε βάσει συμφωνίας συνεργασίας. Στην πράξη όμως έχουμε την εντύπωση ότι είναι παρεμφερή τα καθήκοντα ε, στον τομέα αυτό για την ΕΚΤΕ και για την Eurostat. Ζητάτε παρεμφερή δεδομένα δηλαδή. Θα έχετε μια ε, διαβούλευση εμπειρογνωμόνων ώστε να υπάρξει εναρμόνιση των απαιτήσεων ως προς τις Εθνικές Στατιστικές Αρχές και τις Εθνικές Τράπεζες ώστε να μειωθεί το άχθος που φέρουν ε, οι Εθνικές Αρχές για την εκπόνηση και διαβίβαση στατιστικών ε, στοιχείων. Τώρα, Κάναμε μία πρώτη ανάγνωση στο Κοινοβούλιο για την πρόταση κανονισμού για την ε, παροχή και ποιότητα στατιστικών στοιχείων ε, για τη διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών. Έχετε ε, πληροφορίες σε σχέση με το Συμβούλιο, γιατί καθυστερεί η θέση του Συμβουλίου. Νομίζω ότι μπορώ να είμαι πολύ σύντομο για αυτά που με ρωτήσατε για τις εθνικές ελεγκτικές αρχές και τις διαδικασίες. Να σας εξηγήσω τι έγινε στην Ισπανία. Πήραμε μια τέτοια ελεγκτική έκθεση από έναν, ε, μια περιφερειακή ελεγκτική αρχή στη Βαλένθια, όπως σας είπα, και ε, μας δημιούργησαν ανησυχίε, ήρθαμε σε επαφή με την Εθνική Αρχή, προσπαθήσαμε να το συζητήσουμε μαζί τους, ούτω ώστε να ε, κάνουμε ένα πρώτο απολογισμό των δεδομένων με τη βοήθεια, ξαναλέω, των εθνικών αρχών. Δεν ε, προβλέπεται αυτό από κάποια νομοθετική ρύθμιση. Εμείς ε, στον ιστορικό τρόπο λειτουργίας μας προκρίναμε αυτή τη συνεργασία με τις εθνικές αρχές. Δεν υπάρχει πράξη κατεξουσιοδότηση ή νομοθετική πράξη που προβλέπει ότι συνεργαζόμαστε με εθνικές αρχές. Δεύτερον, για τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ας το διατυπώσω ως εξή. Υπάρχει ένα κεκτημένο, στο πω έτσι, για τι στατιστικές ρυθμίσεις. 200 ομοθετικές πράξεις στο σύνολο περίπου αφορούν και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Είναι έτσι δομημένες αυτές οι πράξεις ώστε τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα να δίνουν, να διαβιβάζουν στατιστικά στοιχεία στην Ένωση και αποφασίζουν τα κράτη-μέλη ποιος κάνει τι ε, ανάμεσα στις αρχές. Βάσει αρχής αποκρουικότητα. Ε, αποφασίζουν ότι η Εθνική Τράπεζα θα διαβιβάσει τα στοιχεία για την, ε, τους λογαριασμούς. Άλλοι αποφασίζουν ότι είναι δουλειά της Εθνικής Στατιστικής Αρχής. Δεν είναι αυτό το θέμα μας όμως θέμα είναι πώς ε, πρέπει να φροντίζουμε ώστε να μην υπάρχει επικάλυψη όταν εκπονούμε νομοθεσία σε επίπεδο ένωσης. Εμείς λέμε, σαν ε, Eurostat, ότι ένας πυλώνας στατιστικών υπάρχει και είναι η νομική βάση 338, το άρθρο 338 Συνθήκης Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε ε, εθνικές τράπεζες ε, που ε, έχουν διοριστεί από τις Εθνικές Στατιστικές Αρχές ως αρμόδιες. Ε, για την διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών MIP είναι εν αναμονή, αν θέλετε, ο φάκελος αυτός, διότι δεν μπορέσαμε να ξεπεράσουμε το πρόβλημα που περιέγραψαν νωρίτερα, όταν μια εθνική τράπεζα αναλαμβάνει τον υπολογισμό ενός εθνικού δίκτυ. Κανονικά θα λέγαμε ότι εμείς ελέγχουμε, η Eurostat ελέγχει αν ε, ε, ε, ευσταθούν τα στοιχεία. Όμως τότε υπάρχει διαφωνία σύγκρουση με την ΕΚΤ. Λέει η ΕΚΤ ότι ακόμη και αν ληφθεί η απόφαση σε εθνικό επίπεδο τότε... Εμείς επειδή αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στην ανεξαρτησία της Εθνικής κεντρική Τράπεζας ε, δεν μπορεί να επέμβει η Eurostat. Υπάρχει ελεγκτικό κενό, ας το πούμε έτσι. Χρειάζεται διμερή συμφωνία ανάμεσα στην Επιτροπή και την ΕΚΤ. Και, συγγνώμη, τη Eurostat διορθώνει ο μιλητής και την ΕΚΤ. Ευχαριστώ. Ε, θα κάνω κι εγώ μια ερώτηση, τελευταία. Πρωτού υποβάλλω την ερώτηση, ε, θερμή έκκληση να συνοηθείτε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξέρετε ότι εμείς ε, ήμασταν διατεθειμένοι να το δεχτούμε. Δεν θεωρούσαμε ότι είναι τόσο σημαντικό το ώστε να ε, παρεμποδίζει όλη τη διαδικασία. Αυτή είναι η έκκληση που ε, σας απευθύνω. Ερώτηση τώρα για την ε, διαδικασία μακροοικονομικών ισορροπιών. Αναφερθήκατε σε διάφορες κατευθυντήριες ε, αρχές ε, για μια πιθανή λύση. Αναρωτιέμαι. Στα πλαίσια της αμοιβαίας εγγύησης ποιότητας, αν κατάλαβα καλά αυτά που είπατε, ενδεχομένως να σημειωθεί ε, πάρα πολύ μεγάλη πρόοδος σύντομα στο Συμβούλιο. Και τρίτον, ορισμένες φορές η <coughs> μέτρηση του διαστρωτικού ελλείμματος είναι κάτι που δύσκολα μπορεί να οριστεί. Και ξέρω ότι βασικά είναι πολιτικό και οικονομικό το ζήτημα, όμως υπάρχουν και στατιστικές επιπτώσεις, δηλαδή από πλευράς μεθοδολογίας, από πλευράς οικονομικής πολιτικής, Θα έπρεπε ίσως να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση, ούτω ώστε να έχουμε αντικειμενικούς ε, τρόπους ε, για να κάνουμε την αξιολόγηση, για να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία για την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Σας ευχαριστώ, λέει ο για τον ε, δίκτυ καταναλωτών δεν νομίζω να ε, είναι θέμα. Το HSCP θα ολοκληρωθεί, ε, μικρή είναι η απόσταση που Και τώρα... Ε, και ε, έχουμε μιλήσει με την, Ευρωπαϊκή Επιτροπή φυσικά και με τη Μελλοντική Προεδρία, την Ολλανδική Προεδρία και το συζητούν εσωτερικά. Και το εξετάζουμε λοιπόν. Το πρόβλημα ποιο ήταν η σύγκρουση ανάμεσα στην ε, ανεξαρτησία τραπεζική και την ανεξαρτησία της στατιστικής υπηρεσίας. Ε, ίσως θα μπορούσαμε να βρούμε ε, μια λύση λογική και που ωφελεί για όλους. Για το διαρθρωτικό έλλειμμα, φυσικά. Μετά την περασμένη φορά που το συζητήσαμε, πραγματικά ερευνήσαμε αυτό το ζήτημα. Όμως καταλήξαμε στο ότι δεν θα έπρεπε να το κάνει αυτό η Γιουροστάτε διότι υπάρχουν δύο ε, πτυχές που δεν είναι δική μας αρμοδιότητα. Πρώτον, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ένα οικονομικό μοντέλο και να αποφασίσουμε σε μία από τις δύο περιπτώσεις θεωρούμε ότι είναι δουλειά της ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ και όχι της ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Ευχαριστώ. Νομίζω καλά θα κάνουμε να ολοκληρώσουμε τις μεταρρυθμίσεις για διάφορους λόγους αλλά και γιατί υπάρχει πλέον αυτός ο δομημένος διάλογος ε, και το είπαν αυτά και συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ λοιπόν που συνεχίζετε αυτόν τον διάλογο και την νομοθετική συνεργασία έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία. Uh, five minutes suspensions and then we, we vote. Δύο λεπτά διάλειμμα. Uh, Συνάδελφοι, ας ε, ξεκινήσουμε την ε, ψηφοφορία. Όπως ξέρετε, ε, εγκρίναμε την ημερήσια διάταξη το πρωί. Αναβλήθηκε η ψηφοφορία για την έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και θα ψηφίσουμε μόνο την έκθεση Βέρνερ Langen για την πολιτική ανταγωνισμού να δοκιμάσουμε λίγο αν δουλεύουν τα μηχανήματα. Άρχεται η ψηφοφορία. Δύο, ένας, λείπουν λοιπόν, ακόμα, ναι, πέρας. Είναι ένας φιλελεύθερος παραπάνω. Ναι, δεν έχει ακόμα κάρτα ψωφορίας. Πόσοι άλλοι φιλελεύθεροι υπάρχουν. Μάλιστα. Ε, δεν το, με την καλή έννοια το λέω. Γιατί δεν μπορούμε αλλιώς να ελέγξουμε. Λοιπόν, ξεκινάει η ψηφοφορία για την έκθεση Βέρνερ Λάγκεν, τροπολογία 42 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 43 υπέρ. Κατά. Δεκτή. Ήμκο 20 υπέρ. Κατά. Να την επαληθεύσουμε. Έρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική α. Να την έχουμε. Αρχικό κείμενο παράγραφος 2. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική α σε δύο μέρη μέρος. Πρώτο υπέρ, κατά εγκρίνεται. Μέρος δεύτερο υπέρ, κατά να την επαληθεύσουμε. έχει την ψηφοφορία. Νομίζω ότι έχει εγκριθεί, αλλά... Πέρας. Εγκρίνεται. Ναι, με μία ψήφο διαφορά. Ωραία. Τροπολογία 48 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 49 υπέρ κατά να απορρίπτεται συμβαστική β υπέρ κατά δεκτή συμβαστική σ υπέρ σε δύο μέρη μέρος πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται μέρος δεύτερο υπέρ κατά εγκρίνεται 167 Μπορούμε να τις ψηφίσουμε όλες μαζί, όχι. Να ψηφίσουμε αυτήν υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 168 υπέρ κατά αποχές δεν βλέπω το EFTD συγγνώμη να την επαληθεύσουμε άρχεται η ψηφοφορία πέρας Απορρίπτεται. Ναι, γιατί υπάρχει άλλος ένας ε, που είναι κατά, οπότε ισοψηφία, οπότε απορρίπτεται. Καλά τα λέω. 169 υπέρ, κατά, τα ίδια και πρέπει να την επαληθεύσουμε. Το ίδιο μου φαίνεται, αλλά... Πέρασε. Η ίδια διαφορά. Λοιπόν, 117 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Μπορείτε να ζητήσετε επαληθευσή. 171 υπέρ. Με συγχωρείτε. Το είπα ότι εγώ από εδώ που βλέπω απορρίπτεται. Είναι σαφές. Αλλά αν θέλετε Λοιπόν, 171 υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. 62 υπέρ. Κατά. εποχέ Δεκτή. 63 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ε, το κόμμα σας. Ε, τι να πω. Λοιπόν, συμβαστική D υπέρ. Κατά. εποχέ εγκρίνεται 71 υπέρ κατά αποχές δεκτή 73 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική ή e υπέρ κατά αποχές δεκτή 81 υπέρ κατά αποχές δεκτή 83 υπέρ κατά αποχές δεκτή να την επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. 83. Πέρας. Α, απορρίπτεται. Τώρα έχετε και την κάρτα ψηφοφορίας. Τροπολογία 84 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγώ είχα άλλη εντύπωση, δεν ξέρω. Λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία. Να το επαληθεύσουμε. Συγγνώμη. Ένας ακόμα δεν έχει ψηφίσει. Πέρας. Και εγκρίνεται. Ναι, 85 ήταν αυτή. 84 υπέρ κατά αποχές συγκρίνεται 86 υπέρ 86 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 87 υπέρ κατά να επαληθεύσουμε την 87 αρχιτή ψηφοφορία πέρασε Απορρίπτεται. 88 υπέρ. Κατά. Να την επαληθεύσουμε άρχη την ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 89 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 90 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 10 της ΙΜΚΟ. Τι θέτε επαλήθευση. Να επαληθεύσουμε την 90 άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. ΙΜΚΟ 10 σε δύο μέρη. Μέρος πρώτο υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Μέρος δεύτερο υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται αλλά να την επαληθεύσουμε. πέρας απορρίπτεται ΙΜΚΟ 15 υπέρ κατά αποχές δεκτή ΙΜΚΟ 19 υπέρ κατά αποχές δεκτή ΙΜΚΟ 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή ΙΜΚΟ 18 υπέρ κατά αποχές δεκτή Ήμκο 22 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ήμκο 23 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ήμκο 25 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική F υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 92 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ήμκο 17 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 93 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 95 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή, είναι τα 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή, τροπολογία 100 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 101 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές δεκτό είναι τα δύο υπέρ κατά αποχές δεκτό 102 υπέρ κατά να το επαληθεύσουμε αρχική ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται 103 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική G σε δύο μέρη, μέρος πρώτο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, μέρος δεύτερο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, συμβαστική H υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, 112 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 113 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, συμβαστική I υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, 119 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 120 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 121 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική J υπέρ Α, σε δύο μέρη μάλιστα μέρος πρώτο της J συμβαστικής υπέρ κατά αποχές δεκτή, μέρος δεύτερο υπέρ, κατά, ναι, μέρος δεύτερο. Το μέρος πρώτο είναι να εξετάσει την κυρίαρχη θέση της Google στην αγορά και μέρος δεύτερο χωρίς, α, με αυτή τη διατύπωση, μάλιστα. Ψηφίσαμε ήδη το πρώτο μέρος όμως. Έπρεπε να το έχω διαβάσει πριν. Λοιπόν, μέρος δεύτερο υπέρ. Κατά άποχες νομίζω πως έχει εγκριθεί αλλά να το επαληθεύσουμε άρχιτη ψηφοφορία και πέρας εγκρίνεται τροπολογία 130 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 132 υπέρ κατά εποχές. Δεν βλέπω χέρια, νομίζω ότι είχε εγκριθεί, αλλά παρακαλώ σηκώστε τα χέρια σας. Παρακαλώ οι συντονιστές, άρχιτε ψηφοφορία. Τουλάχιστον, ναι. Λοιπόν, πέρας. Όχι, όχι εσείς. Από πίσω. Λοιπόν, εγκρίνεται. 134 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 135 σε δύο μέρη μέρος πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται μέρος δεύτερο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 136 υπέρ κατά νομίζω πως απορρίφθηκε αλλά να το επαληθεύσουμε άρχεται η ψηφοφορία Πέρας. Απορρίπτεται. 137 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 138 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να την επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 139 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Ψηφίζεται, απέχουν οι πράσινοι, πέρας, εγκρίθηκε. 141 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 142 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 143 υπέρ, κατά αποχές ε, απορρίπτεται, συμβαστική κάπα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, ε, συμβαστική L υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική M σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα Πρέπει να το διαβάσω. Εντάξει, πρώτο τμήμα χωρίστα τα ε, σε απομονωμένες ή απομακρυσμένες περιοχές και νησιά. Υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 155 υπέρ κατά έλεγχος γιατί δεν βλέπω πέρας απορρίπτεται 156 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι και αυτή απορρίφθηκε υπέρ κατά αποχές. 157 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 158 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται 159 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 161 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 162 υπέρ κατά αποχές αποχές από εγκρίνεται 163 υπέρ κατά ποχές έλεγχος για την 163 άρχεται πέρας απορρίπτεται με μία ψήφο 164 ε, υπέρ κατά αποχές 164 έλεγχος ε, ε, ψηφίστε παρακαλώ πέρασε εγκρίνεται 166 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική εν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 176 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 180 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική όμικρον υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 181 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται μπορείτε να κλείσετε και το συσκευή γιατί βλέπω τα φωτάκια Ήμκο 7 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για την 7 ε, της ΙΜΚΟ Εγκρίνεται. 187 υπέρ κατά έλεγχος για την 187 εγκρίθηκε. Ε, Σημαστική πι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 190 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 192 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 193 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 194 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική Q σε δύο τμήμα το πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές Έλεγχος για το πρώτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Ορίστε. Έγινε λάθος λέτε. Ξαναψηφίζουμε τότε. ούτως ή άλλως εγκρίνεται. Πέρας τώρα. Ναι, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές. Δεν βλέπω να σκόνται τα χέρια, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. Εγκρίνεται. 2.14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική R σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 206 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν βλέπω τους ελεύθερους. Μάλλον υπέρ είστε. Πρέπει να σηκώσετε τα χέρια. Έλεγχος 206. Ε, συγγνώμη, αλλά δεν σηκώνετε τα χέρια. Πέρας, εγκρίθηκε. 208 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 210 υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος. 210. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας, εγκρίθηκε με μία ψήφο διαφορά. 2-12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος και πάλι. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίθηκε. 2-14 υπέρ. Κατά αποχές. Έλεγχος. Πέρας. Εγκρίνεται. Ε, συμβαστική S υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.15 2.25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τάφε σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έλεγχος για το δεύτερο τμήμα άρχη ψηφοφορία πέρας δίκιο είχατε απορρίφθηκε με ισοψηφία τρίτο τμήμα Υπέρ. Εκτός μικροφώνου τα σχόλια δεν ακούνε διερμηνείς. Έχουν δικαίωμα οι συνάδελφοι να μην ψηφίζουν. Τρίτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος στο τρίτο τμήμα. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρασε εγκρίνεται. 2.38 όχι. 207 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική U σε διάφορα τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα. Δεν ξέρω γιατί γράφει πρώτο, λάθος έχουν κάνει. Αφού είναι τρίτο, γιατί το λέει πρώτο. Τέλο πάντων, τρίτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, ε, εγκρίνεται τέταρτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται πέμπτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται έκτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται έβδομο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 2.51 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 2.52 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 2.53 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 2.54 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική έλεγχος για τη 2.54. Νόμιζα ότι ήταν υπέρ το έλεγχο, συγγνώμη. Απορρίπτεται. Συμβαστική Β με προφορική τροπολογία. Ψηφίζουμε για την προφορική τροπολογία. Προχύβη. λέμε αντί για restrict, υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Ό,τι πει η Ελίζα. Πέρασε. Απορρίπτεται. Συμβαστική χωρί την προφορική τροπολογία. Τώρα υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίθηκε. Συμ... Ε, 2.62 υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. 2.63 υπέρ, κατά, έλεγχος η 2.63. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική πι με προφορική τροπολογία των πρασίνων. Α, όχι, διορθώνει ο πρόεδρος W. Για την προφορική, άρα ψηφίζουμε πρώτα. Πρέπει να τη διαβάσω κιόλα. Όχι, είναι μέσα στο κατάλογο. Υπέρ, κατά, έλεγχος, έλεγχος, ψηφίστε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική με την προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική η 2.71 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.72 υπέρ κατά αποχές έλεγχος Νομίζω ε, ότι εγκρίνεται, αλλά έλεγχος. Πέρασα. Εγκρίνεται. 2,74 υπέρ. Κατά. Είναι κατά η πράσινη. Ναι, αλλά όταν είπα κατά, θα σηκώσατε το χέρι. Έλεγχος για να είμαστε σίγουροι. Πέρας. Εγκρίνεται 2,75 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφεται. Συμβαστική X. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2,80 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Είναι 1. Θέλετε όλες μαζί τη Σύντα όχι. Είναι τα 1 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται, είναι τα 5 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται, είναι τα 6 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται, είναι τα 7 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται, είναι τα 8 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται, είναι τα 9 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται, είναι τα 10 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται, είναι τα 11 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική Y υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 96 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 97 υπέρ κατά αποχές δεν βλέπω το EFTD, απορρίπτεται. Θα ψηφίσουμε. Vote is closed. Πέραση της ψηφοφορίας απορρίπτεται. 98 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 99 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Α, ελέγχουμε. Ψηφίστε παρακαλώ. Vote is closed. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Αυτό είναι τμήμα τη συμβαστική. 165 με κατατμήματα ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά. Έλεγχος για το δεύτερο τμήμα. Ε, ψηφίζουμε. Απορρίπτεται. 281 υπέρ. Κατά. Έλεγχος για τη 281. Τέλος. Απορρίπτεται. 282 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Μπορούμε να ψηφίσουμε μπλοκ αν συμφωνείτε. Ωραία. Ψηφίζουμε λοιπόν από τη 83 μέχρι 286. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνονται. 287. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.88 υπέρ κατά. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Τέλος πληροφορίας, ε, ψηφοφορίας εγκρίνεται. Ε, συμβιβαστική Z υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Συμβιβαστική ΑΑ. ΑΑ. Νομίζω εσύ έχετε βάλει. Εγκρίνεται. 299 ε, ελέγχουμε. Vote is closed. A draw. Rejected. Απορρίπτεται. 300 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 301 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 302 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 303 και 304 είναι ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται νομίζω αλλά ας ελέγξουμε. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνονται. 305 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 306 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 307 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, Εκτιμώντα ένα αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, αρχικό κείμενο ε, ε, υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται, τροπολογία 2 υπέρ κατά έλεγχος για την τροπολογία 2 Τέλος ψηφοφορίας.